Buenos días a todos. Se reanuda la sesión de esta comisión y la reanudamos dando la bienvenida a la señora Lisbeth Berhansen, que es la ministra noruega de Pesca y Asuntos Costeros. Καλημέρα Θα ακούσουμε την κυρία Χάνσεν, Υπουργό Αλίας και Παρακτήων Υποθέσεων της Νορβηγίας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που είστε σήμερα εδώ πέρα μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Θα θυμάστε ότι ε, τον Ιούνιο του 2010 είχαμε τη δυνατότητα να σας ε, συναντήσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Ξέρετε ότι επεξεργαζόμαστε την μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής. Χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Σας δίνω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο και θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να προχωρήσω στην ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Ξέρω ότι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Μιλάμε για την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ως Υπουργός λοιπόν Νορβηγίας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ να συνεργάζομαι με όλο τον κλάδο και με τους εκπροσώπους των ε, παρακτήων ε, περιοχών. Η Ελία είναι πάρα πολύ σημαντική για τις παράκτιες κοινότητες και για τους ε, καταναλωτές. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και η Νορβηγία αποτελεί μία από τις χώρες που εισάγει πάρα πολλά προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νορβηγία εξάγει πάρα πολλές ποσότητες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρα πολλές ποσότητες τροφίμων, αλλιευτικών προϊόντων και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σωστό πλαίσιο συνεργασίας μαζί σας. Χρειαζόμαστε ένα ισότιμο επίπεδο συνεργασίας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ισχύουν σωστοί κανονισμοί και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ακούγεται και η φωνή της Νορβηγίας στην θέσπιση αυτών των κανονισμών. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά υφίστανται καταρχάς οι σωστέ συνθήκε ανταγωνισμού. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Έχουμε μεγάλες ροές εμπορικές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νορβηγία και θα πρέπει στο μέλλον να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια καλή χρήση των διαθέσιμων πόρων. Πρέπει να έχουμε στενές σχέσεις, ιδίως όσον αφορά το κατεγάτη και σκατεγάτη. Πρέπει να εργαστούμε επίσης πολύ στενά όσον αφορά τις επικαλυπτόμενες ζώνες εκμετάλλευσης. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια μέσω της συνεργασίας να πετύχουμε μια αύξηση των αποθεμάτων σκουμπριού και έχουν επωφεληθεί βέβαια και οι ελευτικοί μας στόλοι από αυτό. Βλέπουμε τώρα ότι η Ισλανδία και οι νήσες Φαρόες εκμεταλλεύονται το απόθεμα αυτό και θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο γιατί μονομερώς ουσιαστικά εποφελούνται από τις ποσοστώσεις αυτές. Εκμεταλλεύονται λοιπόν ένα 45% των αποθεμάτων αυτών. Πρέπει λοιπόν να πετύχουμε μία ρεαλιστική συμφωνία με όλες τις παράκτιες χώρες. Χρειαζόμαστε μια πραγματική πολιτική βούληση όμως από την πλευρά της Ισλανδίας και των νήσων Φαρών προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και έρχομαι τώρα σε ένα από τα ζητήματα τα οποία σε απασχολούν περισσότερο. Με τα ρύθμιση τη κοινή ελευτική πολιτική. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαραίτητο να ανταποκριθούμε στην πρόταση αυτή. Νομίζω πάντως ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία πλέον προκειμένου να υποφεληθούμε και από την εμπειρία που έχει η χώρα μου, η Νορβηγία. Σίγουρα δεν υπάρχει μια μοναδική μαγική λύση για όλα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν στον τομέα της αλίας. Εν βλέπουμε ότι η καλή διαχείριση των αλευτικών υποθεμάτων συνδέεται με, τις, με τη σωστή διαχείριση των αλευτικών στόλων, καθώς επίσης και με τις απαραίτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που θα μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε ότι τόσο τα λευτικά αποθέματα συνεχίζουν να υπάρχουν, όσο βέβαια και οι θέσεις εργασίας στον τομέα της αλίας. Τη δεκαετία του 1990, η Νορβηγία ουσιαστικά κατάργησε οποιαδήποτε δημόσια υποστήριξη, κρατική υποστήριξη για τον τομέα της αλίας. Ο λόγος που έγινε κάτι τέτοιο είναι ότι οι επιδοτήσεις τελικά αυτές δημιουργούσαν μια κατάσταση πλεονάζουσας αλληλευτικής ικανότητας, η οποία ουσιαστικά απειλούσε τα αλληλευτικά αποθέματα. Λάβαμε λοιπόν αυτή την πολύ σημαντική πολιτική απόφαση και βλέπουμε τώρα ότι ο αλληλευτικός στόλος της Νορβηγίας ουσιαστικά δεν δέχεται επιδοτήσεις. Και επί του παρόντος μπορούμε να πούμε ότι οι Νορβηγοί αλληλείς μπορούν και ζουν πολύ καλά από το επάγγελμά τους. Βέβαια, η πολιτική μείωση της πλεονάζουσας αλληλευτικής ικανότητας ήταν ιδιαίτερα διαφιλονικούμενη. Ήταν σίγουρα μια δύσκολη επίπονη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά επιλέξαμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά βασίζεται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά δηλαδή το σύστημα αυτό των μεταβιβάσιμων αλλιευτικών παραχωρήσεων. Επίσης, έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένου γεωγραφικούς περιορισμούς όσον αφορά τις ζώνες αλλιές και όσον αφορά συγκεκριμένα αλλιευτικά σκάφη. Κατά αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να ελέγχουμε καλύτερα το σύστημα. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι οι παραχωρήσεις αυτές ε, συνδυάζονταν, συγχωνεύονταν. Είδαμε ότι πολλές φορές ε, μειωνόταν από μόνη της η πλεονάζουσα αλλιευτική ικανότητα, χωρίς να χρειάζεται να καταστρέφουμε αλλιευτικά σκάφη. Σήμερα λοιπόν καταφέραμε να επιλύσουμε και ένα ακόμα πρόβλημα. Τη δεκαετία του 90 είχαμε μια πολύ σημαντική μείωση στον αριθμό των αλλιευτικών σκαφών Μειώθηκε επίσης και ο αριθμός των αλλιέων, αλλά δεν μειώθηκε ο αριθμός των αποθεμάτων που αλλιεύονταν. Καταφέραμε λοιπόν να κρατήσουμε ένα σωστό επίπεδο αλλιευτικών αποθεμάτων και να έχουμε τόσο μεγάλο όσο και μικρότερα αλλιευτικά σκάφη. Και το ζήτημα βέβαια της ε, υπερβολικής αλληλευτικής ε, ικανότητας σχετίζεται με το ζήτημα της κερδοφορίας που με τη σειρά του σχετίζεται με το, με το ζήτημα των ε, αποθεμάτων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε έναν πολύ δυναμικό τομέα αλλιές και θα ήθελα να μιλήσω τώρα περισσότερο για τους αλληλευτικούς πόρους. είναι απαραίτητο να έχουμε το απαραίτητο επίπεδο λευτικών αποθεμάτων προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του τομέα αλίας. Και σίγουρα θα πρέπει να εξαλείψουμε τις απορρίψεις. Οι απορρίψεις δεν μπορούν να συνδυαστούν με ένα σωστό σύστημα αλίας. Δεν αρκεί όμως απλώς να προχωρήσουμε σε μια νομική απαγόρευση. Θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα λιεύματα θα μένουν στο σκάφος και δεν θα απορρίπτονται στη θάλασσα. Η απαγόρευση έχει οδηγήσει σε μία σειρά συγκεκριμένων νομικών μέτρων και έχουμε δηλώσει ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχθούμε ότι τρόφιμα μπορούν να απορρίπτονται κατά αυτόν τον τρόπο στη θάλασσα. Η απαγόρευση των απορρίψεων μα επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε κάποιε τεχνολογικέ λύσει προκειμένου να έχουμε μια μεγαλύτερη επιλεκτικότητα στον τομέα τη αλεία. Έχουμε συστήματα προκειμένου να κλείνουν κάποιε ζώνε αλεία. Και ο ίδιο επαγγελματικό κλάδο ε, μα βοηθά αυτή τη στιγμή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα λιεύουμε πάρα πολλά ηχθίδια και γόνου. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι ε, οι αλευτικές ποσοστώσεις θα οδηγούν στη σωστή αλίευση, στην αλίευση των κατάλληλων αλευτικών αποθεμάτων και όχι αυτών που απειλούνται με εξαφάνιση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εγκρίνουμε μέτρα τα οποία στην πράξη θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά. Είναι θετικό λοιπόν να έχουμε μια απαγόρευση απορρίψεων. Η απάντησή μου είναι καταφατική. Δεν σα λέω ότι δεν λαμβάνουν χώρα απορρίψει στην Νορβηγία, ότι τι έχουμε εξαλείψει εντελώ. Έχουμε πάντω ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί σωστά και στα πλαίσια του οποίου οι απορρίψει πια, πια δεν αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Επίσης ήταν καθοριστικό το ότι είχαμε διάλογο και συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Στο Σκαγεράκι έχω εργαστεί πολύ στενά με τους ε, συναδέλφους από την Δανία και τη Σουηδία και καταφέραμε να εγκρίνουμε καταφέραμε να εγκρίνουμε μια κοινή συμφωνία απαγόρευσης των απορρίψεων. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε τις παραδοντικές μας ευθύνες, δεν μπορούμε να μολύνουμε το οικοσύστημα ή να απειλούμε το οικοσύστημα μέσω των απορρίψεων. Θα θέλαμε λοιπόν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι βιώσιμης αλίας σε όλους τους τομείς και νομίζω ότι το Ρίο συνήκωση είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε να παρέχουμε τρόφιμα για έναν όλο και μεγαλύτερο παγκόσμιο πληθυσμό. Το ζήτημα των τροφίμων θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον ένα υγιές λοιπόν οικοσύστημα μπορεί να δώσει και τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις όσον αφορά τα τρόφιμα. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι στην Νορβηγία έχουμε μια πάρα πολύ καλή εμπειρία όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της αλίας. Πρέπει να ληφθούν πολύ καλές δυναμικές αποφάσεις, δύσκολες πολλές φορές αποφάσεις και απαιτείται κατάλληλη ηγεσία. Προχωρήσαμε στι συγκεκριμένε απαγορεύσεις τη δεκαετία του 70, καταργήσαμε ή απαγορεύσαμε τις απορρίψεις τα ζητήματα αυτά από πολιτικής πλευράς ήταν αφιλεγόμενα, έπρεπε όμως οι αποφάσεις πολιτικές αυτές να λάβουν χώρα. Είμαστε λοιπόν σήμερα ικανοποιημένοι που λάβαμε στο παρελθόν τις αποφάσεις αυτές. Προσπάθησα να σας περιγράψω τις ε, σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της αλίας στην Νορβηγία. Δεν σας λέω όμως ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιληθούν ε, τα διάφορα προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Ελπίζω όμω ότι θα καταφέρω να συμβάλλω και εγώ με την εμπειρία μου στην εργασία που κάνετε εσεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε εμεί οι Νορβηγοί να συμβάλλουμε στο να εργαστείτε κι εσεί ε, ομαλά στα πλαίσια τη κοινή ελευτική πολιτική. Η κοινή ελευτική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική για τι παράκτε κοινότητε, για του καταναλωτέ προϊόντων αλληλεία και είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την Νορβηγία. Ελπίζω λοιπόν να συναντήσετε κάθε δυνατή επιτυχία στη μεταρρύθμιση αυτή. Σα ευχαριστώ. <coughs> Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ και πριν να δώσω το λόγο στους βουλευτές που το ζήτησαν θα ήθελα να χαιρετήσω και να καλωσορίσω τον Υπουργό Γεωργίας και Ελιές του κρατηδίου του Βάκλεμπουργκ της Γερμανίας που είναι σήμερα μαζί μας. Και θα δώσω τώρα το λόγο στους βουλευτές που θέλουν να παρέμουν. Πρώτη και καλύτερη κυρία Φράγα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω την παρέμβασή μου σε συγκεκριμένο θέμα σε σχέση με το θέμα των ε, δικαιωμάτων ε, αλληλείας που είναι δυνατόν να μεταφέρονται, αλλά και σε ένα πιο λεπτό ζήτημα, καθώς όπως το γνωρίζει η Υπουργός, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή ε, της ε, σύμβασης του 1920. Όπως γνωρίζετε, η Νορβηγία είναι φυσικά κυρίαρχη στα ύδατά της, όμως λόγω της ισότητας δικαιωμάτων και συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στους αλληλευτικούς πόρους ε, δεσμεύονται όλα τα μέρη και υπήρξε και ένα αντιστάθμισμα το οποίο εδόθη. Ξέρω πως η Νορβηγία έχει πρόβλημα εφαρμογής αυτής της σύμβασης. ιδιαίτερα όσον αφορά τα ψάρια που μεταναστεύουν προς το βορρά και έτσι εξέρχονται της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της ε, Νορβηγίας. Έχουμε δηλαδή εκεί τη δυνατότητα των, α, ε, της παράπλευρης αλίευσης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα. Υπάρχουν δυσκολίες λοιπόν όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της σύμβασης των Παρισίων. Θα ήθελα να μου πει η υπουργό λοιπόν τι σκοπεύει να κάνει, ώστε αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί σωστά, να μην γίνονται διακρίσεις κατά των στόλων μας που επιθυμούν να αλλιεύουν σε αυτά τα ύδατα, να μην γίνονται διακρίσεις και να ε, τηρηθεί πλήρως η σύμβαση των Παρισίων. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε για να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Είναι πολιτικής φύσης, αλλά έχει επιπτώσεις στους αλληλείς διότι υπάρχουν παράπλευρες, ε, παράπλευρα αλλιέματα. Και θα πρέπει να απευθευθεί κάθε διάκριση. Ξέρω ότι η Κομισιόν έχει ασχοληθεί επί μακρόν με αυτό το θέμα αλλά θα ήθελα να μου πείτε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί εμείς ε, είμαστε οι εκπρόσωποι των δικών μας αλλιών που αισθάνονται ότι υπόκειται σε διακρίσεις ε, στα ύδατα αυτά. Να μας πείτε συγκεκριμένα τι σκοπεύετε να κάνετε για να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φράγα. Ο κύριος Ντέιβις. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Υπουργέ. Έχουμε πολλά διδάγματα να αποκομίσουμε από την Νορβηγία. Η εμπειρία σας είναι πολύτιμη. Ε, δύο πράγματα που αναφέρατε, οι απορρίψεις και τα TFC. Και τα δικαιώματα. Ε, Είπαμε ότι αυτά ισχύουν σε διάφορες χώρες όπως η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και ότι θα πρέπει ίσως να τα, κάνουμε, να τα καταστήσουμε υποχρεωτικά. Αλλά όπως είπατε εσείς ε, στην ομιλία σας, ο αριθμός των σκαφών ε, μειώθηκε από 17.000 στις 6 νομίζω είπατε. Και βέβαια μια παρόμοια μείωση γίνεται και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη. Μόνο που ακόμα δεν την έχουμε μετρήσει ακριβώς. Δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, τι συνέβη με τους ε, ψαράδες. Τι έγινε, πήραν ένα εφάπαξ και πήγανε χαροπά σπίτια τους ή απλώς παίρνουν επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι και έπειτα. Τι γίνεται με εκείνα τα, με, με τις ε, αποβάθρες ε, εκφόρτωσης των αλληλευτικών σκαφών είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει και εμείς να αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Τώρα για τις απορρίψεις και άκουσα προηγούμε, ε, πρώην ε, υπαλλήλου ε, στο δημόσιο της Νορβηγίας να λένε ότι οι απορρίψεις τελικά οδήγησε στην αντίστροφη πορεία. Δηλαδή μείωση των παραλιευμάτων και οι απορρίψεις ήταν πολύ σημαντικές για αυτό το αποτέλεσμα. Όταν όμως γίνεται λόγος για την απαγόρευση απορρίψεων στην Ορβηγία, ο κόσμος λέει πως δεν είναι απόλυτο, ότι δεν είναι ε, συνολικό. Γιατί δεν είναι απόλυτο, γιατί, τι κάνουν οι ψαράδες, τα ρίχνουν στη θάλασσα τη νύχτα ή μήπως ε, δεν προσπαθείτε ακριβώς να το επιβάλλετε. Γιατί ο κόσμος λέει ότι αυτή η απαγόρευση δεν είναι 100%, δεν λειτουργεί μάλλον 100% ε, και ότι δεν είναι πραγματική απαγόρευση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, ε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ωστόσο, ήδη τους τελευταίους μήνες είχαμε επαφές με την ε, ε, νορβηγική κυβέρνηση για να δούμε ποια είναι η θέση σας όσον αφορά το βασικό κανονισμό για την πολιτική αλληλείας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις δηλώσεις σας. Ωστόσο θα ήθελα να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις για να εμβαθύνω σε κάποιες ε, πτυχές. Είπατε ότι έχετε σήμερα ένα στόλο πολύ καλά οργανωμένο. Η δυσκολία στην Ευρώπη είναι ότι πολλές χώρες δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν ε, ε, πλεονάζουσες δυνατότητες. Πώς μπορέσατε να αξιολογήσετε και να μετρήσετε τις αλλιευτικές σας ε, δυνατότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς που είναι τα πλεονάσματα, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο καθένας δακτυλοδείχνει τον άλλον και λέει ότι ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και έπειτα έχω μια ερώτηση να υποβάλω στον Chris Davis. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πλεονάζουσε δυνατότητες, ξέρουμε ότι πρέπει να μειωθούν και αυτό με συνέπειε σε ορισμένου αλληλείς που θα χάσουν ε, τα προστοζήν τους. Ε, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να λάβουν κάποια στήριξη όλοι αυτοί. Εσείς τι κάνατε. Ε, φτιάξατε δυνατότητες για να για να απασχοληθούν αλλού όλο αυτός, ο κόσμος ή ε, έχετε δώσει οικονομικές αποζημιώσεις και έπειτα για τις ζώνες όπου απαγορεύεται η αλληλεία. Εσείς είπατε ότι μειώθηκε ο αριθμός των σκαφών αλλά ότι αυξήθηκε ο όγκος των αλληλευμάτων. Πώς καταφέρατε όλα αυτά να τα ελέγξετε, χρησιμοποιήσατε το MSY ή άλλα μέσα που αφορούν την πειθαρχία και τη ρύθμιση τη... των αλλιευμάτων. Και έπειτα, ε, εκεί όπου υπάρχουν ε, ζώνες απαγόρευσης αλλίας, γιατί το κάνατε, επειδή αυτές οι ζώνες είναι προστατευόμενες περιοχές, ας πούμε μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας για τα οικοτόπους και για τις απορρίψεις. Γνωρίζουμε για, τις, ε, για την παράπλευρη αλληλεία ξέρουμε ότι είναι ένα φαινόμενο πολύ διαδεδομένο. Α πούμε στη χώρα μου η αλληλεία γαρίδα είναι, ε, ε, μάλλον σημαίνει πολλά παραλιεύματα, αλλά το θέμα είναι πώς μπορεί να ρυθμιστεί. Εσεί λέγατε ότι δεν δίνονται πλέον επιδοτήσεις, όμως ρωτώ, υπάρχει στήριξη με τεχνική μορφή. Και όσον αφορά την επιστημονική έρευνα, υπάρχει στήριξη από πλευράς της κυβέρνησης? Ποια είναι η κατάστασή σας, γιατί είναι απαραίτητο να συνεχίσει η συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων για να έχουμε ε, μια σωστή αξιολόγηση της κατάστασης. Αυτά είναι τα ερωτήματα που έχω να σας επιβάλλω. Ελπίζω ότι θα μου δώσετε απαντήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Σκούνα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό. Εγώ γεννήθηκα σε απόσταση 55 μέτρων από την παραλία της Βόρειας Θάλασσας. Άρα λοιπόν για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζω ποια είναι η ε, κατάσταση στην Ορβηγία που είναι μια σπουδαία χώρα μια μεγάλη αλληλευτική χώρα και έχει συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία τόσο όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες αλλά και όσον αφορά την βιώσιμη χρήση των, των αλληλευτικών πόρων. Είναι σαφές ότι δεν αρκούν τα ελεγκτικά μέτρα, η παρακολούθηση. Ακόμα και αν καταφέρουμε να παρακολουθούμε κάθε ένα αλληλευτικό σκάφος, γιατί υπάρχει η δυνατότητα παραλίευσης στα δίχτυα ακόμα και όταν κάνει κανείς ε, παθητική αλληλεία. Εσείς λέτε ότι οι ποσοστώσεις είναι χρήσιμες για να δοθούν κίνητρα στους ε, αλληλείς. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει εντοπιστεί μια ποσόστοση για ένα συγκεκριμένο είδος, τι σημαίνει, ότι εκφορτώνονται όλα τα λιεύματα, δηλαδή υπάρχει πλεονάζουσα αλλίευση, εφόσον δεν υπάρχουν πια απορρίψεις. ε, Πομερανία, Δανία και η ε, Νορβηγία μοιράζονται 20.000 τόνους ετησίως του εγκλεφίνου. Τι θα σήμαινε συνεργασία. Συνεργασία θα σήμαινε αμοιβαιότητα ελέγχων και αμοιβαία εμπιστοσύνη στους ελέγχους σημαίνει αυτό πως η νορβηγική εποπτεία θα μπορούσε να επεκταθεί και στα ευρωπαϊκά σκάφη και τα ευρωπαϊκά αλλιεύματα και τούμπαλιν. Προβλέπετε αύξηση λοιπόν της διαφάνειας προς αυτή την κατεύθυνση ή τα νορβηγικά σκάφη λένε ότι το ίμιση το αλλιεύματος του εγκλεφίνου είναι δικιό μας και τα υπόλοιπα δεν τους ενδιαφέρουν. Thank uh, and uh, my words of welcome. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Υπουργό στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Ξέρω ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τον τομέα αλίας της χώρας σας. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες συγκεκριμένε ερωτήσεις που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές για τους αλληλείς που εκπροσωπώ στην ομιλία σας και σας δω συγγνώμη που δεν άκουσα την αρχή της ομιλίας σας. Πάντως έχω την γραπτή εκδοχή της ομιλίας σας και τη διαβάζω. Αναφερθήκατε στην αντιπαράθεση που υπάρχει για το σκουμπρί με τις νήσες Φαρόε και με την Ισλανδία. Ξέρετε ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλέ ανησυχίε στου αλληλεί που εκπροσωπώ, καθώ επίση και στου αλληλεί τη Σκωτία και σε άλλα μέρη επίση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει πολύ συχνά στι συζητήσει τη Επιτροπή μα. Πολλοί από του αλληλεί που εκπροσωπώ ρωτάνε για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρά σε συγκεκριμένε κυρώσει εναντίον αυτών των δύο χωρών. Και με ρωτάνε πότε επιτέλου θα δούμε μια συγκεκριμένη δράση σε σχέση με την Ισλανδία και τις νήσους ε, Φαρόε. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ποια είναι η δική σας η άποψη όσον αφορά το ζήτημα της επιβολής κυρώσεων. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, έλαβαν χώρα πάρα πολλές διαπραγματεύσεις. Πολλές φορές δεν κατέληξαν πουθενά. Βλέπω ότι οι αλληλείς μου πλέον μου ζητάνε να αναλάβουμε δράση. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω σύντομα ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά το ζήτημα ανάκτησης γάδου ιδίως στη Βόρεια Θάλασσα, όσον αφορά το γάδο της Βόρειας Θάλασσας. Πώς θα προχωρήσουμε το ζήτημα αυτό. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας παρατήρησα ότι αναφερθήκατε στην απαγόρευση απόρριψης, απορρίψεων. Εκπροσωπώ λύση από την Ιρλανδία και εμείς έχουμε μία αλία μικρής κλίμακας, μεικτή, παράκτεια είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει απόρριψη, συγγνώμη, απαγόρευση απορρίψεων όταν μιλάμε για συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένα λευτικά αποθέματα. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ποια είναι η δική σας άποψη όσον αφορά τις απορρίψεις για συγκεκριμένα αποθέματα και τις απορρίψεις όταν έχουμε μεικτή αλεία. Το ζήτημα τώρα της πλεονάζουσας λευτικής ικανότητας. Ο στόλος της Βορείου θάλασσας έχει μειωθεί πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Εκεί πέρα που είχαμε πολλές φορές 40-50 σκάφη να λιεύουν ένα συγκεκριμένο είδος, τώρα έχουμε μόνο 2-3. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μία αλία πολύ μικρής κλίμακας, σε αντιπαράθεση με τη βιομηχανική μεγάλη αλία που έχει η Νορβηγία. Θα ήθελα λοιπόν να προστατευτεί αυτή η αλία μικρή κλίμακο και θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η δική σα άποψη και σε σχέση με αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Gracias, señora Κυρία ευχαριστώ πολύ και να χαιρετήσω και εγώ ε, την παρουσία του Υπουργού μαζί μας. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που επέτυχε η Νορβηγία με τη λήψη τέτοιων σκληρών αποφάσεων ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Ήταν μια κρίσιμη στιγμή. Κάποια αποθέματα στην Νορβηγία ήταν ε, στα πρόθυρα της κατάρρευσης και επίσης ε, αναφερθήκατε στην περίπτωση του Εγκλεφίνου ε, στη Βόρεια Θάλασσα. Κατανοώ ε, ότι ήταν πολύ σημαντικό να λάβετε σκληρές αποφάσεις ώστε να δώσετε έναν ορίζοντα ανάκαμψης. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα διδάγματα που μπορεί να αντιλήσει κανεί από το νορβηγικό παράδειγμα και για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Η κυρία Τότσα αναφέρει και σε κάτι που θέλω να θέσω κι εγώ. Αναφέρομαι ε, στα, στην εκφόρτωση των ψαριών και την απαγόρευση απόρριψης, απορρίψεων. Φαίνεται ότι η απαγόρευση απορρίψεων θα είναι πολύ δύσκολη να εφαρμοστεί στην μεικτή αλληλεία. Η Κομισιόν βάζει έναν κατάλογο ε, ειδών που θα τύχουν phasing in με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αν δείτε Σουηδία, Σουηδία-Νορμπηγία και Δανία και τη συνολική απαγόρευση της Καγεράκη, θα δείτε ότι αυτό ήταν παράδειγμα μεικτής αλίας και ε, ε, συγκεκριμένα λοιπόν έχουμε αυτή την εμπειρία που αντίκειται απόλυτα ε, στον τρόπο που βλέπει η Κομισιόν τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει κανείς στο μυαλό του μόνο το γάδο και να γνωρίζει όλα τα άλλα είδη. Ήθελα να ακούσω την άποψη της Υπουργού για το θέμα της απαγόρευσης ε, των απορρίψεων στη Μικτή αλία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαλέσα. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ποσοστώσεις αλίας στην περιοχή Σβέρμπαλτ από την Νορβηγία και την Ρωσία. Παράλληλα βλέπουμε ότι ε, μειώνεται η συμμετοχή τρίτων χωρών στη ζώνη αυτή. Όσον αφορά τις ποσοστώσεις αλίας για την Γρυλανδία, το 2011 είχαμε μια αύξηση που έφτασε μέχρι και τις 18.000. Πολλοί λένε ότι ε, τα αλλιευτικά αποθέματα γάδου και άλλων ειδών στην περιοχή έχουν αυξηθεί. Η Νορβηγία όμως παρόλα αυτά δεν επέτρεψε στην Πολωνία να έχει μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστώσεών της. 140 τόνους μας επέτρεψαν ε, πέρυσι και αυτό δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με τα αρχικά μας σχέδια ή με αυτά τα που είχαμε προβλέψει το 2006. Επίσης δεν καταφέραμε να κάνουμε καν επιστημονικές έρευνες ως Πολωνία στη ζώνη του Σβάρμπαλτ. Το 1920 είχαμε υπογράψει μία συμφωνία που επέτρεπε μία ισότιμη επέμβαση, εκμετάλλευση των υδάτων αυτών ανοιχτά του Βέρμπαλτ. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν τηρεί τη συμφωνία αυτή. Θέτω λοιπόν το ακόλουθο ερώτημα. Δεδομένου ότι ο πληθυσμό των ελευμάτων αυξάνεται σε αυτή τη ζώνη, για ποιο λόγο μειώνουμε για τι τρίτε χώρε τι ποσοστώσει αλλία. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Πρεσέδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Υπουργό για την παρουσία τη. Πραγματικά είναι πολύ καλέ αγαστέ οι θα έλεγα να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Νορβηγία και μα ενδιαφέρει πάρα πολύ η εμπειρία σα. Ρωτώ το εξή λοιπόν. Είπατε ότι εφαρμόζεται το σύστημα <coughs> TFC και ότι το σύστημα αυτό στη χώρα σας ε, έχει δώσει ε, πολύ καλά αποτελέσματα. Ρωτώ λοιπόν ε, κατά πόσον οι ποσοστώσεις αφορούν όλ, όλους τους τόλους και την εραστεχνική αλληλεία και την παράκτη αλληλεία κτλ. ό,τι αφορά τις απορρίψεις. Είπατε ότι είσαστε πολύ ικανοποιημένοι από την απαγόρευση απορρίψεων σε αυτό το τομέα και ρωτώ πώς διαχειρίζεστε εσείς τα προϊόντα που αλλιεύετε και δεν είναι αντικείμενο του κύριου αλλιεύματος, δηλαδή με την εκφόρτωση. Ε, μετά πώς διαχειρίζεστε το αλλιεύμα και έπειτα τι γίνεται με τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων που δουλεύουν σε νορβηγικά σκάφη τα κοινωνικά τους δικαιώματα ε, έχουν αναγνωριστεί επαρκώς. Έχετε να μας πείτε κάποια στοιχεία γι' αυτό. Ευχαριστώ, κύριο ε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σάντζε Πρεσέδο. Και κλείνοντας το γύρο ε, τραπέζι, καθώς υπάρχουν εδώ πολλοί αγορητές και πολλές ερωτήσεις, θέλω να κλείσω όμως αυτό το γύρο για να απαντήσει υπουργό όπως κρίνει ε, σκόπιμο. Tusen takk for det, og takk for mange spørsmål. Spørsmål over et bredt eh, saksfelt. Eh, για όλα αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσω να απαντήσω, αλλά ήταν ευρύτατα τα ερωτήματα. Θα μιλήσω για τις διαρθωτικές αλλαγές καταρχήν και το τι συνέβη με τους ε, ψαράδες που δεν είναι πλέον ψαράδες. Ε, θα πάρω τους γονείς μου ως παράδειγμα. Εγώ προέρχομαι από ένα ζεύγος αλλιέων. Ε, μικρής αλλιείας, ένα σκάφος 10 μέτρα είχαν. Ε, και τελικά εγκατέλειψαν το σκάφο του και ξεκίνησαν μια επιχείρηση υδατοκαλλιέργεια. Αυτό έχουν κάνει πολλοί αλληλεί στην Νορβηγία και έχουμε επίσης περιπτώσεις όπου πολλοί αλληλεί έχουν ε, ενώσει τις δυνάμεις τους για να κάνουν οικονομίε κλίμακας που επιτρέπουν μια καλύτερη απόδοση. Είναι καλύτερο από την άποψη τη ασφάλεια επίση. Επίσης επιτρέψαμε στους αλληλείς που δούλευαν στα μικρά σκάφη να κρατήσουν ένα. Ένα σκάφος χρησιμοποιείται, αυξάνεται η ασφάλειά του και το άλλο μένει στα λιμάνια. Δηλαδή, όπως πολλοί πιστεύουν, η νορβηγική αλληλεία δεν είναι μόνο μεγάλες κλίμακες. Όχι, τα σκάφη στι περιοχέ μας είναι και μικρά αλληλευτικά σκάφη. Έχουμε λοιπόν μοιράσει τις ποσοστώσεις ανάμεσα στα ε, σκάφη παράκτιας αλίες και αλίες στην ανοιχτή θάλασσα. Αυτό σημαίνει πως κάθε σκάφος έχει τελικά την δική του ποσόστοση. Έπειτα, η απαγόρευση-απόρριψης, αν λειτουργήσε ή όχι. Βλέπουμε τα αποτελέσματα γιατί μπορέσαμε να αυξήσουμε τις ποσοστώσεις. Με ρωτήσατε επίσης για το τι θα γινόταν με τους σπόρους μας αν εξακολουθούσαμε να έχουμε 17.000 σκάφη. Φυσικά η απόδοση του κάθε σκάφους, ανά σκάφος, θα είχε μειωθεί. Εμείς ε, βλέπουμε πως η απόδοση από τη στιγμή που ομαδοποιούμε τα σκάφη αυξάνεται. Έτσι, είχαμε, αν είχαμε μάλλον 17.000 σκάφη, αντί για 6, κανένας δεν θα μπορούσε να κερδίσει από αυτή τη δουλειά. Κύριε Ντέιβις, γιατί λένε ότι δεν είναι 100% η απαγόρευση απορρίψεων και ότι ξεκολουθούν να γίνονται απορρίψεις. Κοιτάξτε να δείτε. Στην ε, αλία μας ε, κάνουμε ελέγχους και κάποιες φορές ανακαλύπτουμε απορρίψεις. Ναι, απαγορεύεται, επιβάλλονται κυρώσεις, αλλά ε, ξεκολουθεί να υπάρχει. Πολύ λίγο μεν, αλλά είναι παράνομο, αλλά πρέπει, αλλά πολλές φορές μπορεί να γίνει. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε ακτοφυλακή, η οποία προβαίνει σε ελέγχους. Έχουμε επίσης ηλεκτρονική και ανείχνευση για τα σκάφη μας. Έχουμε ε, το ημερολόγιο του σκάφους, του πλοίου για, τις, ε, για τα αλλιεύματα κάθε φορά. Και πώς γίνεται ο έλεγχος. Όταν υπάρχουν ε, αλλιεύματα τα οποία είναι για συγκεκριμένο είδος, μπορεί εκεί να κάνουμε πιο συγκεκριμένο έλεγχο και ολοκληρωμένο. Φυσικά, όπως σας είπα, μπορεί να υπάρξουν απορρίψεις. Ο στόχος μας όμως είναι, και το μήνυμά μου εδώ, δεν είναι να πούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε για να πετύχουμε 100% απαγόρευση των απορρίψεων και το αποσύστημα να είναι απόλυτα ασφαλισμένο. Μα δεν είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο. Αν φτάσουμε το 96-97% λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει να έχουμε 100% απαγόρευση. Τώρα, οι πλεονάζουσες δυνατότητες. Η κυρία ρόντα έθεσε αυτή την ερώτηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο και πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τις ε, πλεονάζουσε δυνατότητες. Μπορούμε να δούμε ότι στον νορβηγικό στόλο υπάρχουν και σκάφη, τα πιο μικρά σκάφη, τα οποία δεν κερδίζουν πολλά ότι η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ μειωμένη. Δηλαδή, οι ποσοστώσει εκεί είναι πολύ χαμηλέ ώστε να μπορούν να κερδίζουν. Και αυτή είναι μια απάντηση. Εκεί θεωρούμε πω υπάρχει υπερβολική πλεονάζουσα δυνατότητα για τη συγκεκριμένη ομάδα σκαφών. Με αυτόν τον τρόπο μετράμε την αποδοτικότητα. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για μια έκθεση που αφορά τα προϊόντα της θάλασσας και την αλυσίδα παραγωγής για τα προϊόντα της θάλασσας. Φροντίζουμε ώστε αυτή η αλυσίδα να είναι κερδοφόρα για να είναι και βιώσιμη. Επίση, και αυτή μια άλλη ερώτηση, καταργήσαμε τι επιδοτήσει για του αλληλεί. Γιατί? Διότι θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στου αλληλεί να κερδίσουν τη χρήματα με αυτή του τη δραστηριότητα. Αυτό είναι το σημαντικό για μα. Είναι αλήθεια πω έχουμε πετρέλαιο στην Νορβηγία, αλλά παρά τις, τους πόρους αυτούς δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τους αλληλείς που είναι ελληματικές επιχειρήσεις τους γιατί κάτι τέτοιο δεν χρησιμεύει σε τίποτα θέλουμε να μπορούν να ζήσουν από αυτή τη δραστηριότητα με αυτόν τον τρόπο τα βλέπουμε τα πράγματα και πιστεύουμε πως έτσι θα έχουμε και βιωσιμότητα για τον αλληλευτικό τομέα, γεωγραφικοί περιορισμοί. Ή ε, αν δούμε το βορρά της Νορβηγίας, εκεί γίνεται πολύ αλληλεία μικρής κλίμακας. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε εκείνες τις ποσοστώσεις στη Νότια Νορβηγία, γιατί δεν μπορούμε επίσης να τις ανταλλάξουμε ανάμεσα στις, ε, στην αλληλεία μικρής κλίμακας και στην αλληλεία ανοιχτής θάλασσας. Μόνο έτσι μπορούμε να προστατέψουμε την γεωγραφική κατανομή και τους διαφορετικούς μας στόλους. Στο βορρά, όπως σας είπα, υπάρχει πολύ ε, μεγάλο ποσοστό μικρής φαράκτιας αλίες, Έχουμε πολλούς ε, ψαράδες μικρής κλίμακας με σκάφη μικρότερα των 10 μέτρων και πολιτικά λάβαμε μια απόφαση να μην είναι δυνατή η μεταφορά των ποσοστώσεων ανάμεσα στις διάφορες ομάδες. Και έπειτα ακόμα μια ερώτηση της, της κυρίας Ρόντοστ. Το θέμα είναι ότι έχουμε διάφορες ε, ζώνες ε, υδατοκαλλιέργειας, ζώνες παράκτης αλλίες. Πώς κάνουμε λοιπόν και πώς τα διαχειριζόμαστε. Αλλά αυτά έχουμε σχέδια διαχείρισης τα οποία καλύπτουν το σύνολο αυτών των ζωνών. Είναι σχέδια διαχείρισης με συνοχή μεταξύ τους. Φυσικά λαμβάνουμε υπόψη όλες τις δραστηριότητες που γίνονται σε αυτές τις ζώνες, τις ε, δραστηριότητες offshore, τη αλία, την παράκτεια και δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί στην, στο βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας είναι περίπλοκη κατάσταση γιατί έχουμε τις πετρελαϊκές βιομηχανίες που θέλουν να κάνουν περισσότερες γεωτρήσεις, από την άλλη πλευρά θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα συμφέροντα των ε, αλλιών μας. Πρέπει να βρούμε ωστόσο ισορροπία, να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτές τις ε, περιοχές και θέλουμε να έχουμε και επιστημονικά στοιχεία για αυτές τις διάφορες ζώνες για να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε και πώς θα βρούμε την ισορροπία στα σχέδια διαχείρισης. Τι κάνουμε με τα, την, τα παράπλευρα αλλιεύματα, πώς θα διαχειριζόμαστε όλα τα ψάρια τα οποία πιάνονται εκφορτώνονται. Ακόμα και αυτά που δεν είναι τμήμα μιας ποσόστοσης, γιατί είναι πολύ λίγα ή είναι ένα είδος για το οποίο δεν υπάρχουν ποσοστώσεις. Τα περισσότερα από αυτά τα ψάρια θα πάνε στην αγορά, αλλά μπορούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε νυχθιάλευρα. Οι αλληλείς δεν πληρώνονται ε, πέρα από τις ποσοστώσεις ε, που προβλέπονται, αλλά τα ψάρια εκφορτώνονται. Οπότε, Αυτά τα ψάρια δεν είναι και πάρα πολλά. Οι αλληλείς είναι πονηροί. Θα ψαρέψουν τα είδη για τα οποία θα κερδίσουν τα περισσότερα χρήματα. Είναι λογικό κάτι τέτοιο. Όταν απαγορέψαμε τις απορρίψεις, σας, είπα, ε, και σας το είπα ότι έχουν, έχει υπάρξει λόγω αυτού τεχνολογική εξέλιξη. Ε, έχουν περιορίσει τα μάτια των δικτυών, έχουν αναπτύξει συγκεκριμένους μηχανισμούς και μηχανήματα για να ε, προσαρμοστούν στην απαγόρευση των απορρίψεων. Έχουμε επίση έναν κρατικό οργανισμό που ονομάζεται Καινοτομία στην Ορβηγία που μπορεί να συμβάλλει, να δανείσει χρήματα ας πούμε σε κάποια κομμάτια του στόλου για να αγοραστούν νέα μηχανήματα ή για να γίνει έρευνα για ερευνητικού σκοπού. δις νορβηγικών, ε, νορβη, ε, νορβηγικής κορώνας, δηλαδή 200 εκατομμύρια το χρόνο σε ευρώ περίπου, ε, είναι αφιερωμένα στην έρευνα. Και εδώ μιλάμε για έρευνα για τους πόρους αλλά και για την τεχνολογική ανάπτυξη. Το εν τρίτο του δικού μου προπολογισμού πάει στην έρευνα. Η έρευνα είναι κεφαλαιόδοση σημασία αν θέλουμε να έχουμε γνώσεις για τους διάφορους πόρους που υπάρχουν στη διάθεσή μας. και έπειτα υπάρχει και ένα ταμείο έρευνας για όλα τα προϊόντα της θάλασσας. Εκεί ε, το κράτος στήριξε όλους όσους εξάγουν ψά, νορβηγικά ψάρια προς άλλες χώρες όπου πληρώνουν ένα ε, ποσό σε αυτό το ταμείο, το ερευνητικό και το κέντρο αυτό αποφασίζει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα ερευνητικό ανάλογα με τον τομέα που θεωρείται ο πιο σημαντικός. Αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά και θα έλεγα πως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ε, πολλές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες κυρίως, που δεν έχουν όμως τη διάθεσή τους απαραίτητους πόρους για να κάνουν έρευνα. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν πως αυτό το Ταμείο Έρευνας ε, βοηθά πολύ Τώρα, Σβάλμπαρντ. Ο Υπουργό Εξωτερικών μα είναι υπεύθυνο για τη ζώνη αυτή στο πλαίσιο τη κυβέρνηση. Αλλά ό,τι αφορά την αλληλεία, είναι δική μου αρμοδιότητα φυσικά και έχουμε μια, τη διαχείριση για τη ζώνη αυτή και αυτό μέσα στο πλαίσιο του σεβασμού των συμφωνιών που έχουμε συνάψει και στο πλαίσιο της κυριαρχίας που ισχύει για την ζώνη αυτή. Έπειτα υπάρχει μια μεικτή επιτροπή αλληλείας ανάμεσα στην Ρωσία και την Νορβηγία. Ε, για, την, ε, για τον υπόγλωσσο Έχουμε λοιπόν και τη σύμβαση για τον Βορρά που είναι πολύ σημαντική και διαχειριζόμαστε από κενού αυτό το είδος. Έπειτα, μπακαλιάρος. Ο μπακαλιάρος και η αλληλεία του θα πρέπει να συνεχίζεται ακόμα και αν υπάρχει υπόγλωσσος ως είδος. επαληθεύσω μισό λεπτό τα στοιχεία που έχω εδώ μπροστά μου και τις ερωτήσεις. Ο κύριος Κούν ρώτησε για τις ποσοστώσεις. Εν μέρη έχω ήδη απαντήσει. Ο κύριος Κούν ανέφερε όμως επίσης το θέμα του ελέγχου και της συνεργασίας. Έχουμε, κάνουμε έλεγχο για δύο σημεία. Τον έλεγχο των απορρίψεων. Εκεί η εκτοφυλακή προβαίνει σε ελέγχους στα νορβηγικά σκάφη και έτσι ελέγχουμε και τις απορρίψεις. Και όταν πρόκειται για άλλου είδους ε, ελέγχου, έχουμε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την παράνομη αλληλεία. Και έχουμε καταφέρει να σταματήσουμε την αλληλεία στη θάλασσα του Μπάραντς. 100.000 τόνοι αλλιεύονταν τότε και καταφέραμε να το σταματήσουμε αυτό χάρη σε μια καλή συνεργασία. Ένα σημαντικό στοιχείο ήταν η έλεγχη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελέγχουμε τα αλλιεύματα που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί μπορώ να σας πω πως η συνεργασία μας είναι αψεγάδιαστη. Μικτή αλληλεία στη συνέχεια. Είναι μια πρόκληση αυτή σε σχέση με τους αλευτικούς πόρους. Αλλά αν δούμε την περιοχή Σκάγερακ, βλέπουμε πως είναι σημαντικό να έχουμε μία ποσόστοση για κάθε είδος ψαριού που αλλιεύεται ακόμα και σε μεικτή ε, αλίευση και είναι σημαντικό να εκφορτώνονται όλα αυτά τα ψάρια. Όλα τα ψάρια έχουν μια αναξία, εκτός από αυτά που είναι πολύ μικρού μεγέθους, ε, τα οποία όμως δεν θα αλλιευθούν κανονικά χάρη στα επιλεκτικά μηχανήματα που υπάρχουν. Όμως τα ψάρια έχουν όλα μια αναξία και είναι σημαντικό να προβλέπετε μια ποσόστοση που θα αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Ένα παράδειγμα που δεν είναι ίσως το καλύτερο, αλλά μπορεί να σας δείξει τι συμβαίνει. Το μπακαλιάρο στη Νορβηγία είναι ένα από τα πιο σημαντικά είδη. Και θέλουμε η αλληλεία αυτή να γίνεται όσο γίνεται πιο κοντά στις ακτές. Μια συγκεκριμένη περίοδο αλλιεύεται ο μπακαλιάρος και μετά θα συνεχίζεται η αλλιεία της υπόγλωσσας στον φθινόπορο. Είναι λοιπόν λογικό να προσπαθήσουμε να κατανείμουμε καλύτερα τις ποσοστώσεις μέσα στη χρονιά. Υπάρχουν λύσεις. Μπορούμε να ε, συμβάλλουμε στις ε, ποσοστώσεις έχοντας μία συμπληρωματική ε, ποσόστοση Έχουμε δηλαδή υποποσοστώσεις κατά κάποιο τρόπο που μπορούμε να τις κατανείμουμε σε ολόκληρη τη χρονιά. Μπορεί αυτό να λειτουργήσει τόσο για τον μπακαλιάρο όσο και για άλλα είδη. Συχνά έχουμε διάφορα είδη ε, σε κάθε, φορά, σε κάθε αλίευση, αλλά πρέπει να υπάρχουν ποσοστώσεις για κάθε είδος. Μιλήσατε επίσης για αεραστεχνική μικρής κλίμακας αλληλεία. Όπως σας είπα, στην Νορβηγία υπάρχουν πολλά μικρά σκάφη και φυσικά και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα σκάφη. Έχουμε, κάνει έχουμε λάβει διαρθωτικά μέτρα για τους δύο διαφορετικούς τόλους και έχουμε και αυτή την γεωγραφική κατανομή για την οποία ήδη σας μίλησα. Φαντάζομαι ότι θα, υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που ίσως τα ξέχασα, λυπάμαι γι' αυτό. Α, ναι, για το σκουμπρί. Να πω δύο λόγια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το είπα και στην εισήγησή μου. Ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουμε κατασκευάσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ένα πολύ μεγάλο απόθεμα σκουμπριού. Και αυτό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά μπορούμε να προβλέψουμε να υπάρχει με ψηλότερη ε, ποσόστοση με για την Ισλανδία και τις νήσους Φαρόε, αλλά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό με πολύ μεγάλη ακρίβεια, αν και αυτό θα έπρεπε να κάνουμε, γιατί πρόκειται εδώ για την επιβίωση του είδους αυτές τις δύο οικονομικές ζώνες, Ισλανδία και νήσι Φαρόε. Το Ευρωκοινοβούλιο θα ασχοληθεί με την πρόταση της ε, Επιτροπής σε αυτό το πλαίσιο και όσον αφορά τις κυρώσεις κατά τη Ισλανδία και των νήσων Φερόε ε, είδαμε και ότι επιβλήθηκαν απαγορεύσεις εκφόρτωσης στην τελευταία τελευταίες χρονιές. Δηλαδή, η, το σκουμπρί που αλλιεύεται στην Ισλανδία ή στις νήσους Φαρό δεν μπορεί να εκφαρτωθεί στην Νορβηγία. Για, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ισλανδία, γιατί η Ισλανδία είναι και κερδοφο, σημαντική και κερδοφόρος αγορά για την Νορβηγία. Αυτό κοστίζει ακριβά, γιατί έτσι δεν έχει την πρώτη ύλη που χρειάζεται η βιομηχανία. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, πρέπει να δεχτούν τις συνέπειες της κατάστασης αλλά τα ψάρια που αλλιεύονται παράνομα δεν μπορούν να εκφορτώνονται, δεν επιτρέπεται να εκφορτώνονται στην Νορβηγία. Από την πλευρά της Νορβηγίας αυτό σημαίνει πως οι εμπορικές κυρώσεις θα αντιστοιχούν στους κανόνες του ΠΟΕ. Οι αρχές αυτές είναι σημαντικές και πρέπει να εφαρμόζονται. Αλλά όπως σας έλεγα υπάρχει απαγόρευση εκφόρτωσης για τα σκουμπριά. Η Νορβηγία Λιής είναι κάπως απελπισμένης. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό μπορεί αυτό να, κρατήσει χωρίς να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις. Αυτό δεν το γνωρίζουμε και γι' αυτό και φέρουμε ευθύνη. Πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, απλούστατα. Είναι δύσκολο όμως και περίπλοκο. Η Ισλανδία και η νήσι Φερόε φαίνεται να κατοικούν σε άλλο πλανήτη κάποιες φορές. Στην Νορβηγία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καλή συνεργασία. Εγώ θα συναντήσω την κυρία Δαμανάκη λίγο αργότερα σήμερα και θα συζητήσουμε αυτές τις προκλήσεις. Μακάρι να είχαμε τέτοια συνεργασία και με την Ισλανδία και με τις νήσους Φερό, αλλά δυστυχώς δεν την έχουμε. Αυτά είχα να σας πω και ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Υπουργό. Για να κλείσουμε θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες της Επιτροπής στο πρόσωπό σας. Πιστεύω ότι με την εμπειρία σας και με όσα μοιραστήκατε μαζί μας συμβάλλατε στη δική μας σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό ένας εταίρος, ένας φίλος όπως Νορβηγία να μοιράζεται τη δική της εμπειρία από την πολιτική διαχείριση και διαφύλαξη των αλλιευμάτων. Μιλήσατε και εσείς για συμβολή στο δικό μας έργο, στην αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, πραγματικά συμβάλλετε τα μάλα. Κάνουμε και εμείς ε, μία άσκηση πολύ σημαντική. Η αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και πιστεύω ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγίας θα είναι άλλο και πιο στενές και θα έχουμε όλο και πιο κοινού στόχους. Ε, αυτό φαίνεται και από την πολιτική των απορρίψεων και τι μεταβιβάσιμε αλληλευτικέ παραχωρήσει και από άλλες πρακτικές. κλείνοντα κι εσεί είπατε ε, μιλήσετε για το θέμα του σκουμπριού. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και για μας και σας ευχαριστούμε για την προσέγγιση σας. Είναι πολύ σημαντικό από κοινού να ακολουθήσουμε μία πολιτική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να εγγυηθούμε την βιωσιμότητα και την ε, χρηστή διαχείριση αυτού του αλλιεύματος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι και πάντοτε υπολογίζουμε στην ε, καλή συνεργασία μαζί σας. Επίσης ξέρουμε ότι τα νορβικά προϊόντα είναι προϊόντα ποιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αισθάνεστε ότι είστε στο σπίτι σας όταν έρχεστε σε εμά εδώ. Ευχαριστώ. Muy bien, pues despedimos a la ministra. Thanks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 Να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Είμαστε αναμονή ε, του κυρίου Τζοβάνι Λαβία για να συζητήσουμε το θέμα ε, 14 της ημέρης της Εν τω μεταξύ, να δώσω το λόγο στην κυρία Φράγα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά ε, την παρέμβαση της ε, ε, Νορβηγίδας Υπουργού, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο επέδειξε μεγάλη απροθυμία να απαντήσει. Υπάρχει ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και ε, περιέχεται στην συνθήκη των Παρισίων. Υπάρχει ανταλλαγή σημειωμάτων ανάμεσα στην Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βλέπουμε ότι η Νορβηγία συνεχώς παραγνωρίζει το γεγονός ότι έχει προσυπογράψει την ε, συνθήκη των Παρισίων. Είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό χρόνια, είναι πραγματικά περίεργο, καθώς η Νορβηγία αντιμετωπίζει ε, με διακριτική μεταχείριση τον στόλο της ε, Γρυλανδίας και άλλων όμορων χωρών εναντί, μάλλον εις ε, μάλλον υπέρ του νορβηγικού στόλου, συγγνώμη, και ε, είναι μια καθαρά διακριτική στάση. Αυτό το αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίτρανα. Χρόνια τώρα γίνεται αυτό το γεγονός. Ε, λειτουργεί αυτή η κατάσταση βάρος και των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάτι για να επιληθεί το πρόβλημα με την Ορβηγία. Η Νορβηγία, από ό,τι φάνηκε και από τη μη παρέμβαση, δεν ενδιαφέρεται ούτε καν, ούτε ε, μας δίνει κάποιες εξηγήσει. Μάλιστα, κυρία Φράγα. Ναι. Αν συμφωνεί η Επιτροπή, ναι, θα ζητήσουμε εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να καλωσορίσω τον κύριο Τζοβάνι Λαβία για την ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Εισηγητή για τον προπολογισμό 2013. Ήδη έχει εκπονηθεί το σχέδιο ε, έκθεσης για τους γενικούς κανόνες και τον του 2013 που ε, ψηφίστηκε στην ολομέλεια ε, της 17 Μαρτίου. Τώρα είμαστε αναμονή της ε, ψήφισης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 Σα ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Λαβία για την παρουσία του και για τη συνεργασία, την ενισχυμένη που υπάρχει ανάμεσα στην Επιτροπή του την Επιτροπή Προπολογισμού και την Επιτροπή Αλληλεία στο πλαίσιο της συζήτησης περί προπολογισμού για το 2013. Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω την στρατηγική σημασία του τομέα της αλληλείας ε, λόγω της συμβολής του όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική ευημερία των ε, παράκτων πληθυσμών, την ανάπτυξη την ε, τοπική, τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, την αλυσίδα παραγωγής πριν και μετά την αλληλεία, τη συντήρηση των ε, παραδοσιακών ε, εραστεχνικών ε, τρόπων αλίας θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε στο γενικό αυτό επίπεδο, μάλιστα ε, προβλέποντας κάποια συγκεκριμένα μέτρα για το κοινωνικό πλαίσιο και για την απασχόληση. Θα πρέπει δηλαδή συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψουμε όλα τα μέτρα που θα μπορέσουν να επιτρέψουν την ανάκτηση των πόρων, καθώς και τα προγράμματα έρευνας και συνεργασίας ανάμεσα στους επιστήμονες και τους αλληλείς. Το τελευταίο έτος, ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο 2013 ολοκληρώνεται την παραμονή μια σημαντικής μεταρρύθμισης για τον τομέα, η αλία και η θαλάσσια, ο εμπορικός θαλάσσιος τομέας έχουν ανάγκη από στήριξη και από συγκεκριμένε κατευθύνσεις γραμμές από δημοσιονομικής άποψης η μεγάλη πλεονάζουσα δυνατότητα του κοινοτικού στόλου είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με τις ενισχύσεις κοινωνικο-οικονομικού τύπου το 2013 και να στηρίξουμε τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, για παράδειγμα με την ε, τουριστική ελληνία. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην είσοδο των νέων στον τομέα της αλληλείας. Χρειάζεται να στηριχθεί η παράκτεια μικρής κλίμακας αλληλείας, οικογενειακή αλληλεία. Οι μικρομεσαίες στο τομέα της αλληλείας υποφέρουν λόγω της ε, της αύξησης ε, το, του κόστους παραγωγής πράγμα το οποίο έχει άμεση επιπτώσει στα εισοδήματά τους και στην απασχόληση. θα Πρέπει λοιπόν να στηριχθεί ο τοπικός ιστός μιας μικρής αλληλείας που είναι ριζωμένος στις παράκτης κοινότητες. Είναι απαραίτητη, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα, δε της με στήριξη επικτεταμένη και διαρκή στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να στηριχθούν οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες προβλέποντας το νέο ταμείο, το FEMP, που είναι υποσυζήτηση για την ώρα. Ε, χρειάζονται μεγαλύτερες συμβολές ε, για τον εξυγχρονισμό του στόλου, την βελτίωση των στάνταρ ε, επί των σκαφών, της ασφάλειας επί των σκαφών και για την, την βελτίωση των μεθόδων αλληλείας, περιλεκτικότητα των μηχανημάτων, των εξοπλισμών και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να αποφευθούν, να μειωθούν μάλλον οι απορρίψεις των παραλυμάτων στη θάλασσα και ο αντίκτυπος στους θαλάσσιους τους βιοτόπους. Η κοινή αλληλευτική πολιτική καλείται να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 2020 μέσω της ε, κρίσης, της, της ε, μέσω μιας οικονομίας εφιούς, βιώσιμης και με υψηλά επίπεδα απασχόλησης και, και παραγωγικότητας. Γι' αυτό η επιστημονική έρευνα, η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αλευτικού τομέα χρειάζονται χρηματοδότηση σε διαρκή αύξηση. Και αυτή είναι η έκκληση που κάνουμε προς την Κομισιόν και προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστήσω και τον κύριο Λαβία. Συμφωνώ με τα όσα είπε μόλις τώρα η κυρία Φράγκα. Στις 8 Ιουνίου 2012 εγκρίναμε ένα ψήφισμα και είπαμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό κατά 5%. Είπαμε ότι θα γίνει επίσης μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση και ότι αυτό θα επηρεάσει βέβαια και τον τομέα της αλίας και τους ίδιους σαλείς. Πρέπει να δώσουμε τα κονδύλια αυτά στους αλίες. Να σε επιθυμίσω κάτι ακόμα. Η Κροατία σύντομα θα γίνει κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια παράκτια χώρα. Άρα θα λάβουμε πολύ σύντομα και πολλά αιτήματα από την Κροατία. Δεν θα καταφέρουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες με λιγότερα χρήματα. Επιμένω λοιπόν να αυξηθεί ο σχετικός προπολογισμό και να μην μειωθεί. στο εσωτερικό τη Επιτροπή Προπολογισμών υπάρχουν αποκλίνουσε απόψει. Δεν έχουμε ακόμα συντάξει οποιαδήποτε έκθεση για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο Υπάρχει συζήτηση, υπάρχουν αντίθετε θέσει αντιπαραθέσει, γιατί όπω γνωρίζετε πολύ καλά και στο εσωτερικό των διαφόρων πολιτικών ομάδων υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν σημαντική υποδιέρεση με χωριστά δελτία δημοσιονομικά για κάθε πολιτική, ενώ υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μιλήσουν αποκλειστικά για γενικέ στοιχείε χωρί να μπουν στι λεπτομέρειε για τα, αριθμητικά, για τα νούμερα. Όπω ξέρετε, αυτή, σήμερα συζητείται στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, το, το δημοσιονομικό Κοινωνικό Δελτίο για την Γεωργική Πολιτική και για την Πολιτική Συνοχή. Δύο μεγάλα, μεγάλα κονδύλια. Και Στη συζήτηση γίνεται λόγος ε, προφανώ για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 στο Συμβούλιο, αλλά γίνεται λόγος γι' αυτό, αλλά χωρίς νούμερα. Γιατί εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται νούμερα υπάρχουν κάτι χ, άγνωστη χ. Πολύ γενική συζήτηση ακόμα. Άρα λοιπόν θα δούμε μετά από την σημερινή συζήτηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Μπορεί να υπάρξει επιτάχυνση ή αλλιώς επιβράδυνση στον ορισμό του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά είναι σωστό να το ξέρουν και οι συνάδελφοι, ότι από τη στιγμή που το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν εγκριθεί εγκαίρως, αυτό το οποίο θα ισχύσει για την εκτέλεση και βασικά είναι η διοργανική συμφωνία και άρα ο προπολογισμό του 2013, που de facto θα αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο για να λάβει απλά υπόψη το επίπεδο πληθωρισμού. Υπάρχει δηλαδή μια ε, ε, χρονική παράταση του προπολογισμού και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στο 2013 να κάνουμε την καλύτερη δυνατή κατανομή των πόρων γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει αυτός ο προπολογισμό τη βάση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ.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 Thank σας ευχαριστώ από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο για το ζήτημα αυτό. Να σας πω ποιοι είναι οι βασικοί μας στόχοι κατά την προετοιμασία της ε, μεταρρύθμισης αυτής για την περίοδο 2014-2020. Πέντε βασικές αρχές ισχύουν και για τα α, πέντε ταμεία τα οποία προβλέπονται εδώ πέρα. Συμβολή στη στρατηγική 2020, εξοικονόμηση των πόρων προκειμένου να πετύχουμε προσθέμενη αξία, επικέντρωση στα αποτελέσματα, ενίσχυση εταιρικών σχέσεων, απλούστευση και εξορθολόγηση των αποτελεσμάτων. Θα αναφερθώ τώρα σε κάθε ένα σε κάθε μία από τι αρχέ αυτέ, αναφερόμενοι στι βασικέ αρχέ του κανονισμού. Όλε οι κοινοτικέ πολιτικέ και οι πολιτικέ χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλουν προκειμένου να πετυχαίνουμε αποτελέσματα για τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Ουσιαστικά έχουμε 11 θεματικού στόχου όπου θα διοικητευθούν όλες οι επενδύσεις Όλε οι επενδύσει αυτές θα πρέπει να γίνουν μέσω στρατηγικής προσέγγισης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια ενό κοινού στρατηγικού πλαισίου και τα πέντε αυτά ταμεία και θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να χρησιμοποιηθούν με εθνικές εταιρικές σχέσεις. Στη συνέχεια, επενδύσει θα γίνουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και θα πρέπει να δούμε πώς τα έργα τα οποία θα εγκριθούν συμβάλλουν και αυτά στους στόχους στρατηγικής 2020 θα γίνει εξολόγηση εκ των προτέρων προκειμένου να δούμε αν τα έργα αυτά όντως συμβάλλουν στους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν υπάρχουν κάποια προβλήματα γραφειοκρατικά, εθνικά προβλήματα και θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν τα προγράμματα αυτά με, τα, ε, με τις αρχές τα, οι οποίες ισχύουν για την κοινοτική διακυβέρνηση. Δεύτερη τώρα αρχή. Θεματική συγκέντρωση. Επικρίσεις έχουν ακουστεί στο παρελθόν όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Στο μέλλον λοιπόν αποφασίσαμε να, να επικεντρωθεί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που μπορούν να έχουν την υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία και την υψηλότερη δυνατή επιρροή. Θα έχουμε λοιπόν μία κοινή προσέγγιση με κοινέ διατάξεις όσον αφορά τα πέντε αυτά ταμεία για συγκεκριμένους θεματικούς στόχους και θα ισχύουν οι συγκεκριμένοι κανόνες όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση. Τρίτη αρχή. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα. Πρέπει να πετύχουμε τα αποτελέσματα αυτά, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούμε και τα αποτελέσματα αυτά και να υποβάλλονται απαραίτητε αναφορέ. Πρέπει ο Ευρωπαίο φορολογούμενο να γνωρίζει τι επιτυγχάνεται μέσω τη κοινοτική χρηματοδότηση. Ο κανονισμός λοιπόν θέτει και ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Θα αξιολογούνται σε τακτική βάση τα προγράμματα αυτά και θα προβλέπεται επίσης και ένα κίνητρο 5% ανά πρόγραμμα και ανά κράτος μέλος. Θέλουμε επίσης να αξιολογούμε τα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει και μία επιτροπή αξιολόγησης και θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα λειτουργεί η αξιολόγηση αυτή και σε επίπεδο κράτους μέλους. Δίνονται επίση και περισσότερε πληροφορίε στον κανονισμό αταμείων. Αρχή παριθμών 4. Ενδυνάμωση εταιρικών σχέσεων. Από την εμπειρία και τι εξολογήσει μα έχουμε δει ότι ε, οι εταιρικέ σχέσει, οι δυναμικέ εταιρικέ σχέσει είναι πολύ σημαντικέ για την επίτευξη τη Ευρώπη 2020. Θέλουμε να έχουμε μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και θέλουμε, θέλουμε να συμμετέχουν πολλοί εμπλεκόμενοι φορεί. Στο άρθρο 5 του κανονισμού λέμε ακριβώ ότι θέλουμε να έχουμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και εταιρικέ σχέσει. Βλέπουμε ποιοι θα είναι οι εταίροι οι οποίοι θα συμβάλλουν σε όλα τα στάδια τη εφαρμογή, τη χρηματοδότηση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δοντολογικός κώδικα, ιδέα την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει από άλλα θεσμικά όργανα αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συναντιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα όλοι οι εταίροι. Αρχή παριθμών 5. Απλούστευση των, της επίτευξης αποτελεσμάτων η αρχή αυτή διέπει ε, όλες τις αρχές, όλα τα προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέλουμε να μειώσουμε τις δαπάνες στον ε, το γραφειοκρατικό φόρτο και στον, κοινό αυτό κανονισμό προσπαθούμε να εναρμονίσουμε πάρα πολλούς από τους κανόνες που ισχύουν για τα ταμεία αυτά. Κανόνες που έχουν να κάνουν με την ε, εφαρμογή ε, επιτόπου των ταμείων αυτών, την τεχνική αρρωγή, τις ε, λειτουργίες που έχουν να κάνουν με την ε, δημιουργία προστιθέμενης αξίας, ε, αξιολόγηση των ισολογισμών και το καθεξής. Προσπαθούμε λοιπόν στα πλαίσια ενό καονισμού να συγκεράσουμε τους πέντε αυτούς διαφορετικούς καονισμούς που υπήρχαν. Κατά αυτόν τον τρόπο οι δικαιώχοι των ταμείων αυτών δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν πολλούς διαφορετικούς καονισμούς στη διαχείριση αυτών των ταμείων. Θέλουμε επίση να πετύχουμε και ένα εξορθολογισμό μέσω τη γενικότερη αρχή συναλλογικότητα, μέσω τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθου, μέσω τη ε, ε, νομική αρρωγή. Θέλουμε επίση να έχουμε ξεκάθαρου κανόνε ε, όσον αφορά την υποβολή αναφορών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι συνομοθέτε αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούν τον κανονισμό αυτό και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει από όλου εμπλεκόμενου μία υποστήριξη πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Προσβλέπουμε λοιπόν και στη δική σας υποστήριξη προκειμένου να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω προτιμάσει συγκεκριμένη παρουσίαση, γιατί μας ζητήθηκε να μην επισέλθουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Μας είχαν πει ότι θα κάναμε μια γενική συζήτηση για τις γενικέ γενικές διατάξεις. Ο κανονισμός πάντως για τα ταμεία αυτά θέτει συγκεκριμένου κανόνες για το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, το EMFF. Στις γενικές διατάξεις, στο γενικό καονισμό υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που μεταφράζονται σε συγκεκριμένου στόχους όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε συγκεκριμένες προτεραιότητες της Ένωσης για το EMFF και αυτό μπορείτε να το δείτε στο, άρθρο 6 του καονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Είμαι πάντως διαθεσής για να απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις. Oui, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως το εξήγησαν και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις δύο Γενικές Διευθύνσεις, το πολυσέλιδο αυτό έγγραφο το οποίο μας υπευλήθη δεν έχει να κάνει συγκεκριμένα με τον τομέα της αλίας. Πρόκειται για έναν γενικό κανονισμό που περιέχει κοινέ διατάξεις για πέντε ευρωπαϊκά ταμεία. Πρόκειται λοιπόν για ένα γενικό μέσο, για ένα γενικό εργαλείο, για το οποίο εμεί ω Επιτροπή Αλίας δεν χρειάζεται να τοποθετηθούμε. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη θα κάνει τη δουλειά αυτή. Πρέπει λοιπόν να δούμε εμεί εδώ τι ακριβώς πρέπει να πούμε. Δεν θα συζητήσουμε λοιπόν γενικά εμείς για τον κανονισμό αυτό. Ο κύριος Αλάν Καντέκα άλλωστε έχει κάνει μια έκθεση συγκεκριμένη όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Λίας. Εμείς πρέπει να υποβάλουμε μια γνωμοδότηση μέσω της οποίας θα επιφέρουμε κάποιες τροπολογίες και θα πρέπει στόχος μας να είναι στις γενικές αυτές διατάξεις να εντοπίσουμε τι αφορά πιο συγκεκριμένα τον τομέα της αλίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο γενικός αυτός μηχανισμός, ο νέος αυτός γενικός μηχανισμός, δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα, δεν θα πρέπει να τιμωρεί τελικά τον τομέα της αλίας, αλλά θα πρέπει αντίθετα να τον υποστηρίζει και να τον προωθεί. Θα ήθελα παρόλα αυτά να κάνω τρεις σύντομες παρατηρήσεις όσον αφορά τον νέο αυτοκανονισμό, κανονισμό. Τρεις διαπιστώσεις θα ήθελα να κάνω, ουσιαστικά θετικές, όσον αφορά μια πιο θετική μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη βούληση εναρμόνισης, προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη συνέπεια στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τα πέντε αυτά ταμεία. Στο νέο αυτοκανονισμό δεν προβλέπεται μία τομεακή επιχορήγηση, επιδότηση των ταμείων αυτών. Αντίθετα στόχος είναι βάση συγκεκριμένων στόχων να βρεθούν κάποιες κοινέ κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα κινηθούν και επιχορηγήσεις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η βούληση εναρμόνισης, την οποία εγώ κρίνω ιδιαίτερα θετική. Βλέπουμε επίσης και μια γενικότερη βούληση να δημιουργηθούν περισσότερες προϋποθέσεις όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους των κοινοτικών πολιτικών, ιδιαιτέρως όσον αφορά το ζήτημα της βιωσιμότητας των πόρων, όσον αφορά τα κλιματικά ζητήματα και όσον αφορά και το ζήτημα της προστασίας της βιοπικιλότητας. Μια τρίτη παρατήρηση, διαπίστωση θετική, είναι ότι υπάρχει μια βελτίωση και μια ευάνθηση της εδαφικής προσέγγισης, της λεγόμενης περιφερειοποίησης και ενισχύεται ο ρόλος των τοπικών φορέων. Θεωρώ λοιπόν ότι στην πολυσέλιδη αυτή έκθεση τα τρία αυτά σημεία είναι ιδιαίτερα θετικά και κινούνται σε σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει ωστόσο ένα πρόβλημα πολιτικής φύσης, δεν ξέρω αν θα το συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας, είναι όμως σημαντικό και θα συζητηθεί προφανώς στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, αναφέρομαι στο πρόβλημα της ε, μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, άρθρο 21 του κανονισμού. Αυτή η μακροοικονομική αιρεσιμότητα που ουσιαστικά επιβάλλει στις περιφέρειες να συμμορφωθούν με μια πολύ αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα περικοπούν οι α, χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται για τις περιφέρειες αυτές. Αναφέρομαι στο ζήτημα αυτό, μόνο ότι ξέρω ότι δεν θα γίνει συζήτηση στην Επιτροπή αυτή. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Ελίας. Διαβάζοντας την έκθεση αυτή, δεν μπορώ να πω ότι εντόπισα κάποια νέα εμπόδια ή κάποιες οπισθοδρομήσεις ή παναχωρήσεις όσον αφορά τους δικούς μας στόχους. Οι βασικές μεγάλες πέντε αυτές αρχές της νέας έκθεσης ουσιαστικά συνάδουν και είναι ιδιαίτερα θετικές με την εφαρμογή της νέας ελευτικής πολιτικής. Θα ήθελα να κάνω πάλι τρεις συγκεκριμένε παρατηρήσεις, ε, για τις οποίες θα υποβάλω και σχετικές τροπολογίες. Πρώτον, βλέπουμε ότι θέλετε να εφαρμόσετε με μεγαλύτερη ευρύτητα την αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά την έγκριση κονδυλίων. Και ουσιαστικά δημιουργείται εδώ πέρα μεγαλύτερη ελαστικότητα στην αρχή αναλογικότητας προκειμένου να μπορεί να εφαρμόζεται και σε δικαιούχους μεγαλύτερου μεγέθους, ουσιαστικά και μικρότερου μεγέθους. το να αρχίσει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας με τρόπο πιο ελαστικό θα επιτρέψει τελικά σε περισσότερους δικαιούχους να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια που αφορούν την αλία. Τροπολογία επίσης θα επιβάλλω και για το εξή ζήτημα ενίσχυση της δέσμευσης και του ρόλου των τοπικών περιφερειακών αρχών όσον αφορά την χρησιμοποίηση των πόρων, των κονδυλίων. Τρίτη παρατήρηση, θα υποστηρίξετε περισσότερο την εκ των προτέρων ερησιμότητα, δηλαδή οι προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν εκ των προτέρων, προτού χρησιμοποιηθούν κάποια κονδύλια. Κατά αυτόν τον τρόπο το μέσο τη αλίας θα καταφέρει με πιο έντονο τρόπο να πιέσει διάφορες περιφέρειες, περιοχές να συλλέγουν τα απαραίτητα δεδομένα και αυτό με τη σειρά του βέβαια θα ανταποκριθεί καλύτερα στους στόχους της βιωσιμότητας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα λάβετε πολύ σύντομα τις τροπολογίες αυτές. Και βέβαια οι τροπολογίες αυτές έχουν να κάνουν με την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Πατράου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις που δόθηκαν πολύ λεπτομερείς και αρκετά ξεκάθαρες για τα όσα διακυβεύονται. Θα ήθελα να κάνω ωστόσο κάποια σχόλια. Όλα τα πλεονεκτήματα είναι προφανής ε, στην πρόταση που μας υποβάλλατε. Ωστόσο, εγώ έχω κάποιους δισταγμούς. Γιατί όλη η πρόταση που κάνει η Κομισιόν προβλέπει πως οι τοπικές ε, αρχές ε, θα κερδίσουν αρμοδιότητες, ε, ότι η εφαρμογή θα γίνει ανακοινότητα και όχι ανατομέα ή φορέα. Όλα αυτά τα πλανεκτήματα τα βλέπω και είναι σαφή. Όμως η ανησυχία μου αφορά το γεγονός ότι αυτό το μοντέλο λειτουργίας βασίζεται πολύ σε διοικητικούς, τεχνικούς, πολύ πεπειραμένους που καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν τα διάφορα κονδύλια ώστε να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν στο μάξιμουμ. Ε, πώς θα χρησιμοποιήσουν, απαιτείται δηλαδή σύνδεση και συσχέτιση... ανάμεσα στα διάφορα κονδύλια. Άρα, πολύ επαγγελματισμός στο διοικητικό μηχανισμό... και φοβούμαι Ε, πώς θα χρησιμοποιεί, απαιτείται δηλαδή σύνδεση και συσχέτιση ανάμεσα στα διάφορα κονδύλια, άρα πολύ επαγγελματισμός στην, στο διοικητικό μηχανισμό και φοβούμε πως αυτό το ποιοτικό άλμα που είναι υποχρεωτικό για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά τα κονδύλια σε αυτή τη νέα τους μορφή, δεν θα γίνει. Θα μου πείτε είναι ευθύνη των κρατών μελών, αναμφίβολα. Όμως Πιστεύω πως ε, θα πρέπει να γίνει μεγάλο, μια μεγάλη πορεία μέχρι ότου να φτάσουμε να έχουμε τέτοιο διοικητικό μηχανισμό που σωστά να διαχειριστεί όλα αυτά τα κονδύλια. Βλέπω δηλαδή πως αυτό το πρότυπο θα χρησιμεύσει περισσότερο στις βόρειες χώρες που ήδη είναι προσαρμοσμένοι οι διοικητικοί τους μηχανισμοί για τη διαχείριση ε, τέτοιου, τέτοιου είδους ε, κονδυλίων παρά στις υπόλοιπε. Έπειτα, θα πρέπει επίσης αυτές οι συμβάσεις συνεργασίας να γίνουν, να συναυθούν μέχρι το τέλειο του 2013 για προγράμματα τα οποία θα ε, λειτουργήσουν από το 2014 μέχρι το 2020. Γι' αυτό κατ' ουσίαν ο συμβιβασμός ε, που είναι, μάλλον πρόκειται για μια δέσμευση πολύ κοντινή για την κατανομή κονδυλίων που θα χρησιμεύσουν μέχρι το 2020. Δεν έχουμε δηλαδή και πολύ χρόνο για να Έχουμε μια προσαρμογή του διοικητικού μηχανισμού στη νέα χρηματοδότηση για την εκπόνηση προγραμμάτων που να ακολουθούν τις κατευθύνσεις γραμμές όπως αυτές παρουσιάστηκαν για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο βαθμό αυτή τη νέα, τα νέα κονδύλια και όλα αυτά παρουσιάζονται από την Κομισιόν και πρέπει λέει να έχει συναυθεί η σύμβαση μέχρι το τέλος του 2013. Πιστεύω πως ο χρόνος είναι πολύ, το χρονικό διάστημα αυτό είναι πολύ μικρό και ότι αφού πρόκειται για χρηματοδότηση που θα ρέει μέχρι το 2020. Άλλο σημείο ανησυχία και που σχετίζεται πιο συγκεκριμένα με τα θέματα τα δικά μας, της το Ταμείο Αλίες ή, εν πάση περιπτώσει, τώρα των θαλασσίων υποθέσεων και της αλίες. Βλέπω ότι σε ορισμένες χώρες όπου το Υπουργείο είναι ενωμένο με το Υπουργείο Γεωργίας, Φοβόμαστε ότι η γεωργία που είναι ο πιο ισχυρός τομέας σε σχέση με την αλία θα απορροφήσει και τα κονδύλια της αλίας. Το φοβάμαι αυτό για ορισμένα κάτι μέλη όπου όντως υπάρχει αυτού του είδους η υπουργική ε, οργάνωση. όπου δηλαδή οι προτεραιότητες της Γεωργίας θα επισκιάσουν αυτές τις αλίες και άρα θα υπάρξει και μικρότερη, χαμηλότερη απορρόφηση των κονδυλίων. Πέρα από αυτή την ανησυχία, το γεγονός ότι η πρόταση αυτή της, αυτή της Κομισιόν ζητά να έχουμε μια μεθοδολογία λειτουργίας για τη γεωργία και για την αλία που θα είναι ταυτόσιμη. Τώρα δεν ξέρω ακριβώ ποια είναι, δεν μπορώ να σα πω λεπτομέρειε για το ποια είναι αυτή η γραμμή, αλλά, γιατί δεν έχω μπροστά το έγγραφο μπροστά μου. Αλλά σε αυτή τη γραμμή Έχουμε το Ταμείο της Γεωργίας ε, μαζί με το Ταμείο ε, της Αλίας και προτείνεται αυτό το Ταμείο της Αλίας να λειτουργήσει σύμφωνα με τη βάση του μοντέλου της Γεωργίας. Αυτό τι σημαίνει, ότι πάλι η Αλία αποκτά υποδεέστερη θέση σε σχέση με την ε, γεωργία. Αυτή, αυτός ο τρόπος λειτουργίας όμως στον τομέα, τη λειτουργία στον τομέα της γεωργίας δεν χρησιμεύει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια στην Αλία. Θα ήθελα λοιπόν να έχω τη δυνατότητα και να συζητήσω άμεσα με τον εισηγητή, ώστε να μπορέσουμε πιο συγκεκριμένα, με περισσότερες λεπτομέρειες και με βάση τα έγγραφα, να του αναλύσω καλύτερα ποιε είναι οι ανησυχίε μου και οι φόβοι μου, ιδιαίτερα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα κονδύλια στους τομείς στους οποίους απευθύνονται. Να μην επιτραπεί η γεωργία που ήδη έχει τη δική της μορφή, ε, τους δικούς της ρυθμούς λειτουργίας και τρόπους λειτουργίας να απορροφήσει χρήματα τα οποία καταρχήν απευθύνονται στην ε, αλληλεία. Επειδή όμως τώρα η Κομισιόν παρουσιάζει έτσι πιο αλληλένδετα τα ταμεία και πιο συνδεδεμένα μεταξύ τους, ανοίγουν οι πόρτες ώστε να απορροφήσει ο ένας τομέας κονδύλια του Λουνού. Και η ανησυχία μου είναι μήπως έτσι ζημιωθεί η Ελία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίλσον, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι αναπληρωτής στην Επιτροπή Αλίας. Εργάζομαι κυρίως στην Επιτροπή ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία είναι επί της αρμόδια. Μπορώ να σας πω όμως τι συζητάμε εμείς εκεί, σε αυτή την Επιτροπή. Είμαστε υπέρ της πρότασης αυτής. Θεωρούμε ότι είναι καλό να έχουμε κοινού κανόνες για όλα τα ταμεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλη η εργασία που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά θα πρέπει να στοχεύει στο να επιτευχθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι όπως αυτή της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Γίνεται όμως και πολλή συζήτηση για το ποιε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερε συνθήκες που θα πρέπει να ισχύουν για κάθε τομέα συγκεκριμένα στα πλαίσια αυτής της γενικής προσέγγισης. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ζητήματα τα οποία άπτονται περισσότερο της αλίας. Είναι θετικό το ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένου θεματικού τομεί. Νομίζω ότι θα συμβάλλουμε κατά αυτόν τον τρόπο πολύ στην εργασία που γίνεται στην Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η δική σα άποψη, η άποψη τη δική σα Επιτροπή, στο ότι θα πρέπει να περιφερειοποιηθεί η πολιτική αλεία, ότι θα πρέπει δηλαδή να λαμβάνει χώρα πολύ περισσότερο σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό τη ε, υποεξέταση έκθεσης. Euh, euh, euh, πολύ σύντομα. Καταλαβαίνω τι ανησυχίε τη κυρία ε, Πατράου Θα εξετάσω λοιπόν περισσότερο τι ανησυχίε αυτέ και εγώ είμαι ιδιαίτερα διαλλακτικό, είμαι ανοιχτό σε νέε προτάσει, όπω για παράδειγμα για το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω θα πρέπει να το μελετήσουμε αυτό περαιτέρω. Πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Και για την πιθανή αυτή σύγχυση ανάμεσα στη γεωργία και την αλληλεία για την κατανομή των πόρων. Και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εν γέννη όμω, ξέρω πολλέ φορέ ότι ο διάβολο κρύβεται τελικά στι λεπτομέρειε, αλλά εν γέννη πιστεύω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε στην, στον νέο αυτοκαονισμό δεν είναι να δημιουργηθεί σύγχυση ανάμεσα στα ταμεία. Αντίθετα μάλιστα, στόχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό δραστηριότητας και να εξυπηρετούν κοινού στόχους στα ταμεία αυτά. Θα εξετάσω λοιπόν πάντως όλες οι πτυχές του ζητήματος και η ουσιαστική συζήτηση θα επικεντρωθεί στη συνέχεια μέσω της έκθεσης ΚΑΤΕΚ στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Εκεί θα εξετάσουμε τις λεπτομέρειες, αν θέλετε, του ζητήματος Αλίας. Ευχαριστώ. Comenzaríamos, en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 Κατά. Ε, Perdón. Sí. Votamos, votamos la. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα μας ακούτε. Ευχαριστούμε. Τέλο τη ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. ψήφοι υπέρ, ομοφωνία. Ομοφωνία έγκριση. Τώρα μας ακούτε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε. Αρχίζει η ψηφοφορία και πάλι. Από το ατόδος. Ψήφισαν όλοι. 25 ψηφίσατε και εδώ ομοφόνος. Ευχαριστώ πολύ και ε, να ευχηθούμε τα καλύτερα στον κύριο Στίβενσον. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σημείο 12, ληφτικές δυνατότητες. Συγγνώμη, το σημείο 11 είμαστε ακόμη, ψηφίζουμε κατευθείαν για την εξαγωγή τη βιώσιμη αλληλεία και διατήρηση των ηχθιαποθεμάτων. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία με την τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ και την τροπολογία 8. Ο κύριο Γαλαγέρ. Όχι, όχι, ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Την τρία. Από την τρία ξεκινάμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Από τα τόδο, σε Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Τερμίνα. 25. Unanimidad. Seguimos. Votación número 4. Τροπολογία 4. Θα... Άρχεται η ψηφοφορία. Finaliza. Aprobada 23 votos. Ε, εγκρίνεται με 23 ψήφου. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Ομοφόνο εγκρίνεται. Τροπολογία 20 καταπίπτει. Τροπολογία 21 άρχεται η ψηφοφορία. Φιναλίθα. Πέρας. Απροβάδο Ομοφόνος εγκρίνεται. Τροπολογία 6 άρχεται η ψηφοφορία. Finaliza. Πέρας. Εγκρίνεται με 19 υπέρ και 2 κατά. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Φιναλίθα. Πέρας. Ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομοφόνο με 24 ψήφους. Τροπολογία προφορική τώρα. Έχουμε μια προφορική τροπολογία στο άρθρο 4.1 Δέλτα. Κύριε Γκάλετερ, θα είμαι σύντομος σε διαβούλευση με τον Όλικρινσεν των Σοσιαλιστών. Το συζητήσαμε το θέμα και από κοινού υποβάλλουμε αυτή την τροπολογία. Στο κείμενο της Κομισιόν μετά από διαβούλευση με την νομική του Κοινοβουλίου, η τροποποίηση διευρύνει το πεδίο εφαρμογή ε, των κυρώσεων που μπορούν να επιβληθούν σε τρίτε χώρε. Αυτό προτείνουμε. Την έχετε μπροστά σας αυτή την ε, τροπολογία που ουσιαστικά θα αντικαταστήσει τροπολογία 22 και 8. Παρακαλώ, τροπολογία 1, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται ομοφόνος με 25 ψήφους. 22 λοιπόν και οι 8, όπως είπαμε μόλις πριν, καταπίπτουν. Πάμε στην τροπολογία 23, που θα αντικαταστήσει τροπολογία 9. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά. Τροπολογία 10. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομοφόνο με 24 ψήφου. Τροπολογία 24. Ψηφίζουμε. Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 16 ψήφου κατά και 8 υπέρ. Τροπολογία 25. Άρχεται ψηφοφορία. Aprobada. Εγκρίνεται. 11, η 11 καταπίπτει. Τροπολογία της ΔΕΦ... Όχι, διορθώνει ο Πρόεδρος. Καταπίπτει, καταπίπτει και τρο... Ε, εγκρίθηκε 22. Ε, η δεύτερη προφορική τροπολογία, ο κύριος Γκάλγκερ θα πάρει το λόγο και πάλι. Αυτή η τροπολογία, Πρόεδρε, αφορά το άρθρο 6 παράγραφος 3 υπέβαλε την προφορική τροπολογία από κοινού με τον Άλεν Κάντεκ. Το κείμενο της Κομισιόν ζητούμε μια τροποποίησή του, ώστε να συμπεριλάβουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενό μήνα ε, για το κράτος, το εν λόγω που θα πρέπει να απαντήσει στην κοινοποίηση. Θεωρούμε ότι τέσσερις μήνες είναι υπερβολικά μεγάλο διάστημα και ε, κατανοούμε ότι και η Κομισιόν είναι υπέρ του ενό μήνα. Να το υποβάλουμε σε ψηφοφορία την τροπολογία 2, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε Πέρας. Απροβάδα. 17 Λοιπόν, 17 υπέρ, 8 κατά. Πάμε τώρα στην προφορική τροπολογία υπαριθμών 3. Κύριε Γκάλαγκερ. Uh, to... Αυτή η τροπολογία, αυτό το 8-3, είναι νέο σημείο. Υπέβαλε αυτή την ε, νέα τροπολογία μαζί με τον άλλον Κάντακ. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά στην υποχρέωση της Επιτροπής ε, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο την έκθεση αξιολόγησης. Αυτό το προβλέπει ήδη ο κανονισμός 182 του 2011. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μας ακούτε και πάλι τώρα από αυτό το μικρόφωνο. Παρακαλώ, μας κάνετε ένα νόημα να ακούτε τα ελληνικά. Α, ευχαριστώ πολύ. Απροβάδα. Εκρίνεται. Τροπολογία 3. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Rechazada por 14. Ε, καταψηφίζεται, μάλλον απορρίπτεται με 9 ψήφου υπέρ και 13 κατά. Πάμε τώρα στην τροπολογία α, 13 θα την, ψηφίσουμε σε τμήματα. Πρώτα απ' όλα, άρχεται η ψηφοφορία για τη 13. Πέρα. για το πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται Πάμε στο δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Πάμε στην τροπολογία 14. Ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. ΔΕΒ 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Αρχίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση συνολικά όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τέλος το νομοθετικό ψήφισμα ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται ομοφόνος. Ευχαριστούμε και θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Γκάλαγκερ. Α, queda, Λοιπόν, όπως συμφωνήσαμε, μπορούμε Πραγματικά να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Σα καλούμε να εγκρίνετε ε, επισήμως ε, την διαπραγματευτική εντολή προ του ηγητέ. Φαντάζομαι ότι αυτό ε, το εγκρίνεται. Πάμε στο σημείο 12 τη ημερήσιας διάταξη. Αλληλευτικέ δυνατότητε χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται συμφωνία αλληλευτική σύμπραξη με τι Ευρωπαϊκέ Ένωση και τι Δημοκρατίε Μοζαμβίκη. Η κυρία Γκαρθία Ερέρο έχει το λόγο. Εδώ. Perdón, señor presidente. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα απ' όλα σε αυτή τη βασική αρχή της, του επιμερισμού των εξουσιών και της δημοκρατίας. Εδώ ψηφίζουμε μια έκθεση επί της οποίας εγώ εργάστηκα για 24 ώρες και σας ζήτησα να μου υποβάλλετε ερω... προτάσεις. Ε, και από την ΔΕΒΕ και από τον προπολογισμό ε, ζήτησα προτάσεις και θέλω να επισημάνω ότι για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται τρία μείζωνα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, σεβασμός της αλίας, υπό την έννοια της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας επίση να λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα Τη στιγμή που θα υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδου συμφωνίε και πρωτόκολλα οι εργασιακέ σχέσει και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των πληρωμάτων και να γίνεται σεβαστό ο μισθό τους και η συλλογική του σύμβαση με βάση τους κανόνες του ILO Επίσης, αγώνας κατά οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων εργασιακών, φιλετικών ή ε, διακρίσεων ε, κατά του φύλου. Θέματα λοιπόν που είναι πολύ σημαντικά ώστε να μπορεί, θεωρώ, το Κοινοβούλιο πριν λαμβάνει απόφαση και πριν ε, εξετάζει ένα πολιετές πρόγραμμα Θέλω να πω ότι αυτές είναι γενικέ αρχές που πάντοτε οι ειδικοί που εξετάζουν τέτοιου είδου συμφωνίε να εξετάσουν κατά πόσον αυτές οι συμφωνίε λαμβάνουν προ αυτά τα στοιχεία. Μόνο έτσι θα μπορούμε να δούμε αν πρακτικά οι πολιτικές μας εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ώστε να μην καταλήγουμε σε μια συμφωνία όπου επιτρέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράφει ένα πρωτόκολλο αλίευσης σε ε, ξένα ύδατα, αλλά κατά πόσον αυτές οι γενικές αρχές που συζητούμε εδώ και χρόνια και συζητούμε εκ νέου στα πλαίσια της νέας μεταρρύθμισης λαμβάνονται υπόψη. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με άλλα λόγια, να γίνεται σεβαστό το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ε, εισηγήτρια, έχετε δίκιο θα αρκούσε τώρα να μας πείτε ένα ναι ή ένα όχι και να πω ότι έρχεται η ψηφοφορία για την ε, έκθεση αυτή. Πέρας. 18 ψήφοι υπέρ και 3 ε, κατά εγκρίνεται. Παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, έβαλα την κάρτα την πιστοτική μου κάρτα αντί για την ε, κάρτα ψυχοφορίας. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει θέμα ούτως ή άλλως διαφορές. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο ε, το σημείο 16 για την ε, τροποποίηση του κανονισμού 1185-2003 για την αφαίρεση τεριγίων καρχαρία επί του σκάφου. Ήδη έχουμε λάβει πριν από κάποιου μήνε την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ήδη κάνει και θα δούμε σήμερα ε, την έκθεση τη κυρία Πατράου Νέβε, η οποία λαμβάνει και αμέσω το λόγο. Λίγο ησυχία παρακαλώ ώστε να μπορέσει να κάνει την εισήγησή τη η κυρία Πατραονέβες και οι υπόλοιποι να μπορούμε να την ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το έγραφο εργασία. το έχετε όλοι. Ήδη είδε και κάποιο χρονικό διάστημα. Και άρα θα είχατε και το χρόνο να το μελετήσετε και όπως ξέρετε μάλλον εδώ τώρα θα προσπαθήσω να συνοψίσω ποια είναι η δική μου πρόταση και ποια ελπίζω ότι θα είναι η δική σας σε συμβολή έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια πρόταση που να βρει την συνένεση για αυτό το θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα αντιφατικό. Η σημερινή πρόταση της Κομισιόν για την απαγόρευση της κοπής των πτερυγίων των καρχαριών επί των σκαφών υποβάλλεται ως ε, με στόχο να απαγορεύσει τελείως την κοπή πτερυγίων, το φίνιγκ. Ε, και έχω εδώ και ένα σχετικό ανακοινωθέν τύπου από πλευρά τη Επιτρόπου. Ωστόσο, η Επιτροπή ήδη είχε θεσπίσει την απαγόρευση τη κοπή των πτερυγίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003 προβλέποντας όμως κάποιες εξαιρέσεις, εξαιρέσεις όχι για την κοπή πτερυγίων, αλλά για την κοπή των πτεριγιών επί του σκάφους. Ε, το 2005 η Κομισιόν επικύρωσε την ε, ανυπαρξία του Φίνιγκ. Το 2011, ωστόσο, είπε ότι υπάρχουν ε, υποψίες χωρίς όμως να, να υπάρχουν αποδείξεις για τη συνέχιση αυτής της ίδιας πρακτικής. Επίσης, οι ΜΚΟ που στηρίζουν την πρόταση της Επιτροπής δεν μπόρεσαν να μας δώσουν στοιχεία αποδείξεις ότι συνεχίζεται η κοπή των πτυριγίων. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αυτό το οποίο είναι το διακύβευμα δεν είναι ακριβώς η πρακτική του φίνιγκ, για το οποίο δεν υπάρχουν αποδείξεις. Αυτό που το θέμα είναι η απλή δυνατότητα διατύπωσης ε, υποψιών που προκύπτουν από ένα ανεπαρκές επίπεδο ελέγχου που να είναι σε θέση να εξαλείψει όλες τις ε, υποψίες. Αυτό το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή είναι τα... Ε, μάλλον αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι στοιχεία και αυτά δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Από τα στοιχεία προκύπτουν δύο γραμμές πιθανής ενημέρωσης και ανανέωσης. Πρώτον, πρώτη γραμμή δράση. Το να πετήσουμε η Κομισιόν, σύμφωνα με την αρχή της λήψης τεχνικών μέτρων και πολιτικών μέτρων, με επιστημονική βάση, να ανακαλέσει την πρότασή της, μέχρι ότου να έχει στοιχεία τα οποία να την αιτιολογούν ε, να προτείνει νομοθεσία με βάση υποψίες, υποψίες οι οποίες όμως δεν στηρίζονται σε στοιχεία είναι ένα πολύ σοβαρό ε, ζήτημα. Πολύ σοβαρό ζήτημα ε, για, που θα μπορούσε να γενικευθεί με αυτή την αρχή της ε, δράσης επί αβάσιμων στοιχείων. Πρόκειται για υποψίες, αμφιβολίες, έλλειψη εμπιστοσύνης, που πάντως δεν είναι επιβεβαιωμένες. Αυτή τη στιγμή που δουλεύουμε για την μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής και όπου συμφωνούμε με την Κομισιόν και έχουμε ομοφωνία μεταξύ μας ότι η μελλοντική μεταρρυθμισμένη κοινή ελευθερική πολιτική θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία, θα ήταν ε, παράλογο και θα αποτελούσε και σοβαρό προηγούμενο το να δεχτούμε αυτήν την αρχή, ε, η οποία δεν μπορεί να σταθεί την αρχή δηλαδή των, της υποψίας, της ύπαρξης μάλλον υποψιών ή αμφιβολιών. Αυτή λοιπόν η ανάκληση η κατα... που εγώ έχω εδώ ορίσει ως πρώτη δυνατότητα δράσης συνοδεύεται ως από την αιτιολόγηση της έλλειψης ε, μελέτης αντικτύπου από πλευρά της Κομισιόν που προκύπτει από την ίδια της την πρόταση γιατί εμείς ακόμα μια φορά συμφωνούμε ομόφωνα με την Κομισιόν ότι η μελλοντική μεταρρυθμισμένη κοινή ελευτική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει αυτή η μελέτη κοινωνικο-οικονομικού αντικτύπου. Σας είπα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές δυνατότητες δράσης. Την πρώτη σας την παρουσίασα και σας ε, παρουσιάζω και τη δεύτερη. Η δεύτερη δυνατότητα είναι να παρέμβουμε σε ένα επίπεδο όπου τοποθετείται πραγματικά το πρόβλημα. Δηλαδή, την απάλληψη των υποψιών. Όντως, από τη στιγμή που το πραγματικό πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε είναι ο έλεγχος ε, της αλληλείας καρχαρία και ανεπάρκεια ελέγχου και όχι η ύπαρξη του ή όχι του φίνιγκ, η δική μας δράση θα πρέπει άμεσα να παρέμβει όσον αφορά τις διαδικασίες ελέγχου στα σκάφη. Πώς μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε τον έλεγχο. Εγώ θα έλεγα και προτείνω υποχρεωτική ταυτόχρονη εκφόρτωση στο ίδιο λιμάνι των σωμάτων, των κορμών και των ε, πτερυγίων ώστε να μπορούμε άμεσα να δούμε ποιο πτερίγιο αντιστοιχεί σε ποιο κορμό. Η θέσπιση ενός ε, καθεστώτος ελέγχου αναπερίπτωση και όχι με προειδοποίηση. Δηλαδή, όπως έγινε ήδη με άλλα είδη. Αυτή η ενίσχυση του ελέγχου πώς μπορεί να γίνει χωρίς αύξηση της χρηματοδότησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξωτερική συνεργασία από πλευρά των πλειοκτητών, ε, με έναν οργανισμό, επίσημο οργανισμό ε, επιστοποίησης, όπως ε, για παράδειγμα το γραφείο βέρετας, ώστε να προβαίνει αυτό στους ελέγχους. Με άλλα λόγια, ήδη αυτό έχει δοκιμαστεί και κοστίζει 8 με 10.000 δολάρια ανασκάφο και, ανα, και Άλλη πρόταση είναι η ε, ανάθεση της ευθύνη στον ίδιο τον πλειοκτήτη με ορισμό ενό εκπροσώπου μιας ΜΚΟ, την οποία ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ο οποίος ε, παρατηρητής μπαρκάρει ως παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε μία μαρτυρία για, πρώτον για το γεγονός ότι δεν γίνεται το φίνινγκ, δεύτερον διότι διαφορετικά οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικές. Θα πρέπει λοιπόν τις δύο πτυχές αυτές να τις, να τις εξετάσουμε ε, χωριστά. Ο Ευρωπαϊκός Στόλος δεν κάνει φίνη, γιατί θα ήταν η οικονομική αυτοκτονία. Εδώ και 15 χρόνια που αναπτύχθηκε η αγορά για το κρέας του Καρχαρία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έτσι ώστε κάθε ζώο το οποίο αλλιεύεται να είναι αντικείμενο εκμετάλλευση. Ε, σήμερα θα σας πω ότι ακόμα και το σηκώτη του Καρχαρία πωλείται προς ένα ευρώ το κιλό. Ακόμα και η πώληση του κορμού μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρο. Είναι σαν το σχήρος αυτή τη στιγμή ο Καρχαρίας. Εκμεταλλεύονται κάθε κομμάτι του σώματος του ψαριού αυτού. Άρα λοιπόν ο Ευρωπαϊκός θόλος θα ζημιωνόταν αν εγκρινόταν η πρόταση της Επιτρόπου. Έχουν υπολογιστεί ανά σκάφος ψυγείο και ανά αλευτική περίοδο και προκύπτει η ζημιά από την επιπλέον εργασία, τις υπερορίες, τη μείωση του χώρου που είναι απαραίτητος και σε μια εκτίμηση που έχει γίνει, που είναι μια χαμηλή εκτίμηση, έφτασα στις 33,7% μείωση του κέρδους. Μείωση σχεδόν 34% του κέρδους. σημαίνει 9,5 ε, εκατομμύρια ευρώ ζημιά ανά για τον Πορτοκαλικό και ισπανικό στόλο. Αυτά είναι τα στοιχεία στα οποία φτάσαμε σε συνεργασία με τον κλάδο. Και αν η Κομισιόν έχει κατατύχει άλλου είδους υπολογισμού στη διαθεσή της, να μας τους παρουσιάσει, παρακαλώ. Και αν παρευχήν, παρελπίδα προσχωρήσει με αυτή την ε, πρόταση της Οικομισιόν θα πρέπει να μας παρουσιάσει την μελέτη κοινωνικο-οικονομικού αντικτύπου. Θα μπορούσαμε ίσως να προβλέψουμε δε και μια τρίτη γραμμή δράσης ε, συμπληρωματική με τη δεύτερη, δηλαδή την δυνατότητα εξαίρεσης. Μέσω της μελλοντική δυνατότητας εφαρμογής της πρότασης της Κομισιόν, κάτι τέτοιο θα ζημίωνε κυρίως τον στόλο των σκαφών ψυγείων και θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει στον περιορισμό της κοπής των πτεργίων ε, επί του σκάφους μόνο στα σκάφη ψυγεία και να εξαιρεθεί ο στόλος ε, του νοπού ψαριού. Έτσι θα μειωνόταν ο αριθμό των σκαφών τον οποίο θα πρέπει να γίνει ο έλεγχο και θα συμβάλαμε μαζί με τις προηγούμενες προτάσεις στην μείωση των υποψιών για φίνινγκ ε, σε μηδενικό επίπεδο. Τέλος. Θα αξίζει τον κόπο να σα πω ότι το 90% των καρχαριών που αλλιεύεται από τον Ευρωπαϊκό Στόλο είναι ενό συγκεκριμένου είδου. Αυτό το είδος οριμάζει πρώιμα, δηλαδή στα 4 με 5 έτη ζωής του και έχει μια σημαντική βιολογική παραγωγικότητα με μέσο όρο 35 έμβρια ετησίως μπορώντας να φτάσει, και μάλιστα μπορεί να φτάσει και στα 80 έμβρια ετησίως. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και που μας τα έδωσε η ΑΕΚΑΤ αλλά και διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με τη συντήρηση του, του, του θαλασσίου περιβάλλοντος επι, επιβεβαιώνει ότι το αλίευμα αυτό, αυτό το είδος δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι πάνω από, τις, ε, από το MSY. Υπογραμμίζω μάλιστα ότι οι επιστήμονες γενικά, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, Λένε λοιπόν πως έχουν ε, καλές σχέσεις με τους πλειοκτήτες τους επιτρέπουν ε, κάθε φορά που το επιθυμούν να ανεβαίνουν στην, ε, στα σκάφη και μάλιστα μου είπαν ότι με τη συνεργασία των πλειοκτηκτών, με τη δική τους καλή θέληση, έχουν ξεκινήσει την καταγραφή ενός μητρώου. Έχει περισσότερες μάλιστα λεπτομέρειες στο Μητρό αυτό από αυτές που προβλέπει το, ο νόμος και με διαβεβαίωσαν ότι έχουν κάθε δυνατότητα πρόσβαση στα σκάφη. Και αυτό για να σας πω ότι οι σχέσεις αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν. Και κάθε φορά έχουμε ακόμα περισσότερα στοιχεία για την αλληλεία του Καρχαρία. Χάρη στους επιστήμονες με τους οποίους ήρθα σε επαφή. Αυτό που εγώ προτείνω λοιπόν και πάντοτε με βάση την αρχή ότι αυτό που εδώ διακυβεύεται δεν είναι το φίνινγκ αλλά η ενίσχυση του ελέγχου για να εξαλειφθούν υποψίες περί φίνινγκ θα ήθελα να προτείνω να υπάρξει περιορισμός των εξαιρέσεων στα πλοία ψυγεία μόνο, να υπάρξει έλεγχος ε, που θα επιβαρύνει τους πλειοκτήτες όχι αναπερίπτωση αλλά τυχαία, με τυχαίο δείγμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, αυτές τις ε, ζημιές που θα υποστεί ο στόλος, γιατί η μεταρρύθμιση ε, θα σημάνει λιγότερους ψαράδες, λιγότερα σκάφη και φυσικά και οικονομική ζημιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Έξι αγορητέ έχω στο κατάλογό μου. Θα σα παρακολουθήσω να είστε σύντομοι για να, προλάβουμε. να προλάβουμε. Ο κύριο Αρσένη πρώτα απ' όλα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με την κυρία Πατρά Ονέβες, συναντηθήκαμε αρκετές φορές. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση που να βασίζεται στην κοινή λογική, σε δεδομένα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή μια συναισθηματικά φορτισμένη συζήτηση. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα εκφράσω και τις παρατηρήσεις μου, τις έχω εκφράσει και σε άλλες συνεδριάσεις βέβαια. Δεν θα πω κάτι το ιδιαίτερα καινούριο. Εξετάσαμε και με τη βοήθεια των βοηθών μου όλα τα σημεία της έκθεσης του εισηγητή. Εξετάσαμε επίσης και στο παρελθόν την αρνητική οικονομική επίπτωση που εκφράζεται από την εισηγήτρια πολύ στεναρά στο δεύτερο έγγραφο εργασίας. Συμφωνώ με την μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μελέτη η οποία δεν δείχνει ουσιαστικά ότι υπάρχει μια σημαντική οικονομική επίπτωση στον επαγγελματικό αυτό κλάδο, δηλαδή επίπτωση η οποία προέρχεται από τα μέτρα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα δεύτερο τώρα ζήτημα, η υγιεινή, η απειλή υγιεινής, κίνδυνη υγιεινής. Τι προκύπτει δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί αν ε, διατηρήσουμε στο σκάφος ε, όλα τα πτερίγια τα οποία είναι προσκολλημένα στο σφάγιο. Ξέρετε ότι ε, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα εντόστια, ούτε μπορούμε να κόψουμε το κεφάλι, δηλαδή είναι τμήματα τα οποία σαπίζουν πολύ γρήγορα. Επομένως, αν διατηρήσουμε τα πτερίγια προσκολλημένα στο σφάγιο, δεν φαίνεται να υπάρχει μια επίπτωση. Το ζήτημα της ασφάλειας τώρα. Δηλαδή πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι τα πτερίγια όταν είναι κατεψυγμένα δεν ισχύει ενα τέτοιος κίνδυνος αν κόψουμε εν μέρη τα πτερίγια και τα διπλώσουμε στο πλάι του κορμού του ζώου, στο πλάι του σφαγίου δηλαδή. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε και να εξοικονομήσουμε χώρο και καταστούμε τελικά το σφαγείο πολύ πιο ασφαλές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το ίδιο ισχύει και για τα αλλιεύματα που έχουμε στη θάλασσα, Μάλλον αν διπλώσουμε τα πτερίγια δεν τίθεται και το ζήτημα του χώρου, της έλλειψης χώρου. Όσον αφορά τώρα την απουσία δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε κάποιες περιπτώσεις παραβίασης του κανονισμού και βλέπουμε ότι και με τις υφιστάμενες διαδικασίες η παρακολούθηση, η εποπτεία είναι πολύ δύσκολη. Επομένως δεν μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε πιο μικρές περιπτώσεις παραβίασης. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Ένα πράγμα επιτρέψτε μου να πω κύριε Πρόεδρε. Δεν λέμε αυτή τη στιγμή κάτι καινούριο. Ουσιαστικά λέμε αυτό που οι διεθνείς εταίροι μας και οι φορείς της αγοράς μας λένε. Αυτό κάνουν και άλλες χώρες όπως ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, αυτό κάνουν και χώρες της ΙΚΑΤ και χώρες όπως η Κολομβία και άλλες. Κύριε Αρσένη, εγώ να σας δώσω πολύ προστερό χρόνο αν μπορούσα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ε, πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Το θέμα είναι πραγματικά ο κύριο Τρομέδα έχει πάρει το λόγο. Ξέρετε, το θέμα αυτό ε, είναι σαφές ή δεχόμεθα ή όχι την πρόταση της Κομισιόν. Τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ξεκάθαρα. Είναι σαφές ότι είναι μας αν εγκρίνουμε αυτή την πρόταση, διότι το πρόβλημα του ελέγχου θα καταστεί μικρότερο πρόβλημα, γιατί θα είναι απλούστερος ο έλεγχος. Η προσέγγιση επιστημονική θα μπορεί να εφαρμοστεί πολύ καλύτερα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και επίσης θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρακτική του φίνινγκ από όλα τα έθνη που συνεργάζονται με τους Ευρωπαϊκούς Στόλους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, οικονομικός πώς, αν θέλετε, θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα κέρδη για τον κλάδο, γιατί αυξάνει, αν θέλετε, η αξία του σφάγιου. Λοιπόν, περισσότερος έλεγχος και ε, μια πιο επιστημονική προσέγγιση μας επιτρέπει αυτή η πρόταση. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις συστάσεις ώστε να καταργήσουμε αυτή την παρέκκληση. Γιατί πρώτον, τα στοιχεία μας λένε ότι είναι η καλύτερη επιλογή και δεύτερον γιατί ακόμα και τα ε, άλλα κράτη που κάνουν αυτού του είδους ε, την αλία την κάνουν τόσο άλλως. Ήταν περίεργο λοιπόν να προσπαθούμε να, να δίνουμε μαθήματα σε κράτη-μέλη οργανισμών ότι πρέπει να είναι ε, υπεύθυνα. Είμαστε τελευταίοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει βούληση ο πλευράς εισηγήτριας για κάποιον συμβιβασμό. Αλλά νομίζω τα πράγματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα από ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Εγώ υπερασπίζομαι τη θέση όπως φαίνεται, ε, μάλλον όπως την έχουμε διατυπώσει στο παρελθόν. Πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν, πρέπει να σταματήσει ε, οπωσδήποτε αυτή η παρέκκληση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα κονδύλια για τον έλεγχο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ο καλύτερος ε, έλεγχος και η καλύτερη επιστημονική προσέγγιση είναι κάτι διαρθρωτικό. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο της μεταρρύθμισης. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απλά τα πράγματα να υπερψηφίσουμε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατανοώ τη θέση συγγητρίας, αλλά εγώ πιστεύω ότι το αντίθετο είναι πιο εύκολο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαβάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Ρωμέδα. Πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο ήδη είχε συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στην εμπορία καρχαρία. Επομένως δεν μπορούμε εμείς να βγούμε προς τα έξω και να προτείνουμε χαμηλότερα πρότυπα. Ενώ υπάρχουν χώρες όπως το Εκουαδόρ και η Ταϊβάν που έχουν υψηλότερα πρότυπα από ότι εμείς και ουσιαστικά εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες πολιτικές για την προστασία του είδους αυτού. Η συλλογή τώρα περισσότερων δεδομένων ποιες είναι οι πραγματικές δαπάνες προκειμένου να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα σταματήσει η πρακτική του φίνινγκ. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που εμπλέκονται, ακόμα και αναπτυσσόμενες χώρες. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε συγκεκριμένο αριθμό πτερυγίων που θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα σφαγεία. Πολλές φορές από τα πτερυγία Μάλλον, όταν κόβουμε τα πτερίγια και πολλές φορές αφαιρούμε ακόμα και το κεφάλι ή το δέρμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, γιατί είδος καρχαρία ε, πρόκειται. Υπάρχουν χώρες όπως ο Καναδάς που έχουν ένα ποσοστό αντιστοίχησης 5%. Πάντω η κατάσταση σε διεθνέ επίπεδο είναι ιδιαίτερα βέβαιη και θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζητάμε περισσότερα δεδομένα όταν έχουμε τις απαντήσεις διαθέσιμες τελικά. Η συγγήτρια μας λέει ότι θα πρέπει να έχουμε και τα πτερίγια προσκολλημένα πάνω στο σφάγιο και ότι θα πρέπει να εκφορτώνονται στον ίδιο λιμένα. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα πάντως του κλάδου. Ο κλάδος πολλές φορές μας λέει ότι τα πτερίγια μπορούν να πηγαίνουν σε έναν λιμένα, το δέρμα σε κάποιον άλλον. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε κανέναν ψάχνοντα να βρούμε μια συμβαστική λύση. Νομίζω ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κρατήσουμε τα πτερίγια προσκολλημένα στο σφάγιο. Κυρία Φράγα, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, για κάποιες αναφορές που ακούστηκαν από τους προλαλήσαντες, θα ήθελα να πω το εξής. Το πρόβλημα που αφορά τους ευρωπαϊκούς στόλους είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι αντιμετωπίζουν άλλοι στόλοι. Γιατί το πρόβλημα αφορά τους στόλους που ε, προέρχονται στην κατάψυξη το προϊόντος, ενώ εσείς συγκρίνατε με άλλους τρίτους στόλους που μεταφέρουν μόνο νοπό προϊόν δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Το πρόβλημα αυτό αφορά μόνο στόλους που κάνουν κατάψη προϊόντος. Και να πω ότι ε, σε μια χώρα από που αναφέρατε, μόνο μόνο ένα σκάφος ε, προβαίνει στην κατάψη του προϊόντος. Οπότε δεν θεωρώ σωστή τη σύγκριση. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα ελέγχου. Η εισηγήτρια πολύ ωραία μας εξήγησε τη διάθεση του στόλου που κάνει την κατάψευση να προβαίνει στην εκφόρτωση από κοινού στο ίδιο λιμάνι. Συμφωνεί, συμφωνεί λοιπόν ο στόλος να εκφορτώνει από κοινού πτερίγια και κορμού ζώου και να αναθέσει τον έλεγχο σε οργανισμό πιστοποίηση όπως οι και κτλ ενώ το κόστος είναι τόσο υψηλό, οπότε κατανοείται ότι αν η ίδια η βιομηχανία είναι διαθέσιμη να το κάνει αυτό, τότε ποιος είναι ο οικονομικός αντίκτυπος που αντιμετωπίσει. Το βασικό ζήτημα λοιπόν που τίθεται εδώ και αυτή είναι η επικριτική μου στάση ανά της Κομισιόν είναι ότι κάνει μια πρόταση Κομισιόν που αφορά τον Καρχάρια και μια ευαίσθητη κατηγορία αυτή, αλλά δεν έχει τηρήσει την υποχρέωσή της να κάνει μια ορθή μελέτη αντικτύπου. Λαμβάνοντα υπόψη τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο ε, ε, μιας απόφαση. Αυτό δεν το έκανε η Κομισιόν. Δεν τήρησε μια μεγάλη υποχρέωσή τη. Εργαζόμαστε εδώ και μήνε με τον κλάδο και με τις κυβερνήσεις για να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει αυτό το μέτρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα θυμάστε, την τελευταία φορά που ήταν εδώ, δεν ήταν σε θέση καν να μα πει πόσα σκάφη θα πληγούν από αυτό το μέτρο. Αυτό, αυτό είναι ο ψόγο που έχουν να, ε, να απευθύνω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι στο μέλλον. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε καταλήξει σε προτάσεις ε, με συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία επαληθεύει και ο κλάδος και η τα κράτη-μέλη, οι κυβερνήσεις. Ρωτώ λοιπόν, ποιος θα αυτά τα στοιχεία η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβαδίζει με τις γενικές αρχές που θέτει η ίδια, ότι δηλαδή έχει κάνει τον κατάλληλο κοινωνικό αντίκτυπο. Πρώτα, ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός για την απαγόρευση της ε, φέρεσης πτερυγίων, είχα πει και εγώ ότι θα πρέπει πτερύγια και σφάγιο να εκφορτώνονται στον ίδιο λιμένα μαζί. Είχε απορριφθεί αυτό τότε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή πανέρχεται τώρα και κάνει την ίδια ακριβώ πρόταση. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό, Γιατί έχουν πλέον υποψίε ότι οι βέλτιστε πρακτικέ που μα είπαν ότι ίσχυαν στο παρελθόν τελικά δεν ισχύουν. Συμφωνώ λοιπόν με την εισηγήτρια που σαν καλή δικηγόρος έχει χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα επιχειρήματα με τα οποία είμαι σύμφωνος και πιστεύω ότι αν χρειαστεί ποτέ να πάω στο δικαστήριο, σε σένα θα απευθυνθώ, Μαρία. Νομίζω όμως ότι αντέστρεψες κάπως την ε, αρχή της πρόληψης. Αντί να πεις ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα και επομένως θα πρέπει να, να ισχύει η αρχή πρόληψης, είπες ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα και δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα από αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι να έχουμε τα δεδομένα αυτά. Ακούσαμε όμως ότι αλλού στον κόσμο υπάρχουν ελευτικοί στόλοι οι οποίοι εκφορτώνουν μαζί πτερίγια και σφάγια. Η ανησυχία μου όμω, οι ανησυχίε παραμένουν και υπάρχουν κάποιε υποψίε ότι υπάρχουν κάποια κενά στον νόμο τα οποία ορισμένα εκμεταλλεύονται. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω αναφερόμενο στην έκθεση της ε, εισηγήτρια, η οποία σε ένα σημείο λέει ότι οι περισσότεροι καρχαρίες εκφορτώνονται σε τροπικές τρίτες χώρες με υψηλές θερμοκρασίες και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ε, συνθήκες υγιεινής προκειμένου να αποθηκευθούν τα σφάγια αυτά. Και όντως αυτό μπορεί να ισχύει, ότι όντως δεν υπάρχουν απαραίτητες συνθήκες υγιεινής στις χώρες αυτές. Έχουν όμως ε, και τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να καταχωρούν όλα αυτά τα στοιχεία σε Μητρώα. Κυρία Στίβενσον, για να κλείσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οφείλω να πω στη Μαρία ότι έκανε βεβαίως ε, πολύ καλές προσπάθειες, αν σε επαφή με όλους μας. Και εγώ ως εισηγητής την συγχαίρω για αυτή ε, τη στάση. Όμως, και πάλι εδώ, έχουμε να κάνουμε με το Καρχαρία το Blue Shark το που είναι το 80% των αλλιευμάτων καρχαρία στα ύδατά μας και είναι, έχει διχαρτιστεί ως ευάλωτο είδος για την ε, Μεσόγειο, έτσι δεν είναι. Ε, ε, Mako, which Το επίσης, είναι 10% και αυτό είναι ευάλωτο. Βλέπουμε λοιπόν και τι συμβαίνει στο αν Πάει κανείς ε, στην αγορά. Τι διαθεσιμότητα ε, προϊόντος υπάρχει. Στο βίγκο λοιπόν πώς καταλήγει τόσο μεγάλο εμπόρευμα ε, γλαυκοκαρχαρία. Εσύ η ίδια ε, μας είπες Μαρία ότι κατά κύριο λόγο έχουμε να κάνουμε με σκάφη που καταψύχουν το προϊόν. Αλλά εγώ θέλω να σα υπενθυμίσω ότι έχουμε και πολλές άδειε που δεν έχουν κοινοποιηθεί. Και την τελευταία φορά που το συζητήσαμε το θέμα με την Κομισιόν, τι μας είπε. 120 περίπου είναι οι άδειε που ε, έκαναν αίτηση παρέκκλησης από τον κανονισμό. Άρα οι υποψίες μας πηγαίνουν πολύ παραπέρα. Για να γίνονται τόσες αιτήσει παρέκκλησης, τι σημαίνει αυτό. Για να μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμμόρφωση από όλα τα κράτη-μέλη. Και ο πιο εύκολος τρόπος για να αποφύγουμε ε, δυσανάλογο βάρος για τα κράτη-μέλη πρέπει να εγγυηθούν τη συμμόρφωση είναι να κάνουν εκφόρτωση του Καρχαρία ε, χωρίς να του έχουν κοπεί τα πτερίγια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πατράου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπόθηκε εξ αρχής ότι θα κάνουμε αντικειμενικό και νυφάλαιο διάλογο. Εγώ συμφωνώ ότι αυτό έγινε, αλλά δεν ήταν πάντοτε σοβαρός ο διάλογος. Θα ήθελα να ήταν και σοβαρότερος. Το λέω αυτό γιατί κάποια από τα πράγματα που ακούστηκαν αυτομάτως αναιρούνται λόγω των στοιχείων. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι ο διάλογος δεν ήταν πάντοτε σοβαρός. Για παράδειγμα, το να λέει κανείς ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα στοιχεία από αυτά που ήδη έχουμε, πώς μπορεί κανείς να το λέει αυτό. Χρειαζόμαστε πάντοτε περισσότερα στοιχεία. Πάντοτε και άλλοι μάλιστα είπαν ότι χρειαζόμαστε στοιχεία. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει εδώ. Έχουμε κάποια στοιχεία και χρειαζόμαστε και περισσότερα. Και γι' αυτό μην μου λέτε ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα στοιχεία. Μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα στοιχεία για τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που δεν τα έχουμε. Και εδώ έχουμε τη δέσμευση ότι οι αποφάσεις μας εδώ σε αυτή την Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό αντίκτυπο. Εμείς ήδη έχουμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση εδώ και πολύ καιρό και θα συνεχίσουμε να το λαμβάνουμε υπόψη για την επόμενη μεταρρύθμιση. Ας είμαστε λοιπόν συνεπείς. Και όταν επίσης λέτε κόστος, ότι αυτό de facto θα σημαίνει παραπάνω κόστος. Εγώ σας παρουσίασα δύο λύσεις και σας απέδειξα ότι δεν θα σημαίνουν αυτές οι κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς μου λέτε ναι θα κοστίσει όλο αυτό. Ε, δύο, δύο προτάσεις δράσης σας έδωσα που σας απέδειξα ότι δεν θα επιφέρουν ε, κόστος. Και μετά μου είπατε ότι η βιομηχανία, ο κλάδος δεν θα, δεν θα συμφωνήσει. Μα ε, συμφωνεί ήδη. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με τον κλάδο. Ζητάνε ενίσχυση του ελέγχου. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Επιμένω, κανείς ακόμα δεν μας έδωσε μια απόδειξη για φίνινγκ από τον Ευρωπαϊκό Στόλο. Ούτε μια απόδειξη. Λένε ότι υπάρχουν υποψίες. Μπορεί να υπάρχουν υποψίες συνέχεια πώς θα δουλέψουμε στο επίπεδο των υποψιών, ενισχύοντας τον έλεγχο. Δεν μπορούμε εδώ να μιλάμε για κόστος, λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε, έχετε δύο προτάσεις για ενίσχυση του ελέγχου χωρίς επιπλέον κόστος. Και μάλιστα οδηγισμένες από αυτές τις λύσεις ήδη έχουν δοκιμαστεί. Με τον τόνο. Δεν μπορώ λοιπόν να αντιληφθώ την έλλειψη ε, ε, την έλλειψη θες, ε, ανοιχτού πνεύματος του πλευρά των συναδέλφων για τις προτάσεις τις οποίες σας υπέβαλα εδώ. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις που αντιποκρίνονται στο πρόβλημα. Δεν λέω ότι είναι η πιο απλή. Η πιο απλή μπορεί να μην λειτουργήσει υπάρχουν ορισμένοι που αναζητούν τις απλούστερες δυνατές λύσεις για να αποφεύγουν την πολλή δουλειά. Όχι, εγώ δεν αναζητώ τις πιο απλές λύσεις, ε, αναζητώ τις πιο κατάλληλες λύσεις. Είπαμε λοιπόν, αναπερίπτωση έλεγχο, τον οποίο θα πληρώνει ο ίδιος ο στόλος. Άλλη λύση ε, της ίδιας της Επιτροπής είναι να ορίσει εκπροσώπους των ΜΚΟ που θα ε, βρίσκονται στα σκάφη. Και με αυτές τις λύσεις μου λέτε ακόμα ότι θα κοστίσει ο έλεγχος ο παραπανήσιος. Ε, δεν καταλαβαίνω ειλικρινά. Έπειτα λέτε ότι ο στόλος θα κερδίσει με αυτή τη θέση. Μα ποιοι είστε εσείς που λέτε ότι ο στόλος είναι αυτός που θα κερδίσει, όταν ο ίδιος ο στόλος έχει κάνει τους λογαριασμούς και μας λέει ότι θα υποστήσει μια της τάξης των 1,5 εκατομμυρίων ανά σκάφος. Έχετε άλλα νούμερα. Ωραία, δείξτε τα μου και μετά θα δουλέψουμε με βάση αυτά τα νούμερα, τα δικά σας. Σας παρουσίασα λοιπόν νέες ε, λύσεις, νέες προοπτικές και ειλικρινά υπολόγιζα πως θα είχατε αρκετά ανοιχτό μυαλό για αυτές τις νέες λύσεις που λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή, πιο αποτελεσματικός έλεγχος τόσο στα ευρωπαϊκά λιμάνια όσο και εκτός αυτών χωρίς επιπλέον κόστος. Και μην τυχόν έρθετε και μου πείτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την αντιστοιχία ανάμεσα στα πτερίγια και τα σώματα των καρχαριών, όταν όλα φυλάσσονται επί των σκαφών, οι ίδιοι οι πλειοκτήτες δεν έχουν πρόβλημα να είναι παρόν διαρκώς ένας εκπρόσωπος των ΜΚΟ και να βλέπει ακριβώς τι γίνεται πάνω στο σκάφος. Επίσης, μην μου πείτε πως δεν υπάρχει ζημιά όσον αφορά το θέμα του χώρου όταν έχουμε υπολογίσει ότι έχουμε ένα ε, μειωμένο χώρο κατά 10%. Όταν λέτε πως δεν υπάρχει αντίκτυπος για τη βιομηχανία, δεν είναι αλήθεια, γιατί τα στοιχεία μας το αποδεικνύουν και δεν έχουμε άλλα στοιχεία που να λένε ότι όχι, δεν υπάρχει κανένας αντίκτυπος. Επίσης, μου λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα ελέγχου. Οι προτάσεις που σας υπέβαλα εγώ αποδεικνύουν πως είναι δυνατόν να ελέγξουμε ε, καλύτερα με απόλυτο τρόπο, χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα και χωρίς επιπλέον κόστος. Τι ακόμα που να αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε, διαπιστώσαμε λόγω ε, τη συζήτηση, γιατί υπήρξε και κάποιος διάλογος, ότι κάποιες φορές ε, υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στον στόλο νοπού ψαριού και τον στόλο των σκαφών ψυγείων, αλλά και πάλι σας επαναλαμβάνω ότι αυτό αφορά τον στόλο των σκαφών ψυγείων. Εκεί ο άλλος στόλος, ο υπόλοιπος στόλος του οπού ψαριού δεν επηρεάζεται από αυτές τις ε, εξαιρέσεις. Και φυσικά ο αριθμός των αδειών θα μειωνόταν καθώς πρόκειται μόνο για τα ψυγεία. Και όταν ε, γίνεται λόγος για την αρχή της προφύλαξης και εδώ ο συνάδελφος και φίλος Ντέβις που έλεγε ότι μπορεί να είμαι καλή δικηγόρος, θα το σκεφτώ όταν θα ανακυκλωθώ και θα αλλάξω επάγγελμα. Και μου είπατε ότι δεν χρησιμοποίησα καλά την αρχή της προφύλαξης, γιατί όντως ε, η αρχή της προφύλαξης λέει ότι δεν πρέπει να ενεργήσουμε από τη στιγμή που δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να ενεργήσουμε. Αυτό, ε, αυτή είναι η αρχή της προφύλαξης. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και για περιβαλλοντικά ζητήματα το ότι δεν θέλουμε να υπάρξει παραπάνω πίεση στα αποθέματα από τη στιγμή που δεν έχουμε στοιχεία στη διάθεσή μας που λένε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να ξεπερνάμε το MSY. Εδώ όμως αυτό που ξέρουμε για τις καρχαρίες είναι το 90% του ε, είδους είναι, είναι πάνω από το MSY, πολύ παραπάνω από ότι πολλά άλλα είδη και στον Ατλαντικό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να σας πω επίσης ότι ήρθα σε επαφή με επιστήμονες και στη συνέκρινα στοιχεία της ICAT και της ΕΝ και τελικά είδαμε ότι τα πρότυπα, τα στοιχεία επί των οποίων ε, λειτουργεί το ΣΕΝ δεν είναι ε, κατάλληλα σύμφωνα με ορισμένους ε, επιστήμονες. Ενώ εμείς συνεργαζόμαστε με την το που έχει κατάλληλα πρότυπα για κάθε ένα από τα είδη ψαριών. Ενώ το ΣΕΝ έχει κάποια πρότυπα τα οποία δεν ταιριάζουν για ορισμένα είδη όπως τα, οι καρχαρίες. Επίσης δεν είναι τα ίδια πρότυπα που ισχύουν στον Ατλαντικό και στον ε, Ειρηνικό. Ο καρχαρίας του ωκεανού ε, είναι ένα είδος το οποίο είναι ιδιαίτερα γόνιμο και αναπτύσσεται ταχύτατα ε, οριμάζει στα 5 με 6 έτη ηλικίες και μπορεί να, έχει, να φέρει 35 έμβρια. Οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει επί τόπου δείχνουν ότι είναι σχετικά μικρή η ε, παρακμή αυτού του αποθέματος. Είναι η εκτίμηση του 2009 του IOCN. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αν θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Παρακλείω να είστε σύντομο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα να σχολιάσω κάποια από όσα ακούστηκαν για τη μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν και ποιες είναι πληροφορίες βάσει των οποίων κάναμε την πρότασή μας. Είχαμε μια ανοιχτή διαβούλευση που κράτησε αρκετό καιρό, μήνες, και λάβαμε πολλές αξιόλογες πληροφορίες και από το κλάδο, τον ισπανικό και τον πορτογαλικό κλάδο. Λάβαμε πολλά αριθμητικά στοιχεία, μακροσκελής, λεπτομερείς ε, ε, προτάσεις, χωρίς όμως να μπαίνουν στις λεπτομέρειες που ακούσαμε σήμερα για την εκτιμόμενη ε, ζημία που ανέφερε η κυρία Πατράων Νέβες. Ε, μόλις σήμερα ακούω αυτά τα στοιχεία είχε ο κλάδο να, ε, να στείλει αυτά τα στοιχεία στην Κομισιόν, αλλά μόλι σήμερα τα ακούμε. Σε ό,τι αφορά τα νοπά και κατευσυγμένα αλλιεύματα και τις άδειε που συνδέονται με τα σκάφη ψυγεία και τα σκάφη μεταφέρουν από προϊόν, να πω τα τελευταία χρόνια, οι, οι άδειε αφορούν τα σκάφη ψυγεία. Οπότε, αντί να κάνουμε μια σχετική διάταξη, γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα ουσιαστικά στην κατάσταση, αυτοί που αλλιεύουν νοπό καρχαρία δεν έχουν τις ίδιες άδειες. Οι άδειες, επαναλαμβάνω, που χορηγώ τελευταία χρόνια φορούν τα σκάφη ψυχία. Δεν αλλάζει τίποτα λοιπόν στο status quo σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Συμφωνούμε, πιστεύω όλοι, ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος και θα πρέπει να ενισχυθεί ο απλούστερος και φθηνότερος τρόπος ελέγχου θα μπορεί να υπάρχει όταν τα πτερίγια παραμένουν πάνω στον κορμό του Καρχαρία. Λιγότερος κόσμος, λιγότεροι εμπειρογνώμονες, λιγότερος χρόνος. Αυτή είναι η ιδανική λύση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και αρκετό χρόνο. Να σταματήσω καλύτερα εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε για αυτό το σημείο. Πάμε στο επόμενο σημείο ε, και κλεισμένων των θυρών το πρώτο μέρο, οπότε παρακαλώ όσοι δεν έχουν την ειδική άδεια να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Τα επόμενα 10 λεπτά, εγώ στα τελευταία μάλλον 10 λεπτά λέει ο Πρόεδρος, πάλι η συνεδρίαση γίνεται ε, δημόσια. Λοιπόν, κατανοείτε ποιοι επιτρέπεται να μείνουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κλεισμού των θυρών. Τα μέλη, η γραμματεία και οι συντονιστές και παρακαλώ ησυχία. Στο πρώτο λοιπόν μέρος και κλεισμού των θυρών έχουμε